Um, Καλημέρα συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε με το σημείο 1 που είναι η έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στην ημερησία διάταξη. Σήμερα το πρωί έχουμε ένα σημείο 11α, σχέδιο έκθεσης για το υπόμνημα κατανόησης ε, όσον αφορά την ε, επιχειρησιακή ετοιμότητα και χρήση των IT ε, ε, στον χώρο της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Εάν δεν υπάρχουν, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να σας πω εξ αρχής ότι δεν έχουμε κροατικά και μαλτέζικα στην διερμηνία. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες καλύπτονται. Επίσης ότι στις 11 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έγκριση πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων 28 και 29 Νοεμβρίου 16, 5 Δεκεμβρίου του 2016. Αν δεν υπάρχουν σχόλια και αντιρρήσεις εγκρίνονται και τα πρακτικά και επομένως φτάνουμε στο σημείο 4 και στο σημείο 5 ε, παρουσίαση του, των ε, τριμερών διαλόγων όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τα δύο αυτά θέματα. Ο κύριος ε, της, κύριος Δίας Ντεμέρα, έχει δουλέψει πάρα πολύ έτσι ώστε να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες όσο γίνεται πιο γρήγορα και του δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο. Κύριε Δίας Δεμέρα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξ αρχής όμως θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου με τον Βρετανικό λαό και με τις Βρετανικές αρχές σε σχέση με την τρομακτική επίθεση του προηγουμένου Σαββάτου στο Λονδίνο. Και βεβαίως, και βεβαίως να εκφράσω την ε, βαθιά μου λύπη για, τον, ε, για την βραδύτητα με την οποία αναγνώρισαν ε, την, ε, και ε, έδωσαν στους οικείους του ε, την σωρό του, σύμβα, του συμπατριώτη μου. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Όπως και τα υπόλοιπα θύματα βέβαια. Όσον αφορά το θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και είναι γεγραμμένο στη μερίσια διάταξη, ήθελα να πληροφορήσω τα μέλη της Επιτροπής μας ότι Πραγματοποιήσαμε τρεις πολιτικούς τριμερείς διαλόγους και ο τέταρτος ε, θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα. Είχαμε δέκα τεχνικές συνεδριάσεις, ε, καθώς επίσης και διάφορες άτυπες συνεδριάσεις. Σήμερα το πρωί, μάλιστα, ακόμα μία τεχνική τέτοια συνεδρία, άτυπη τέτοια συνεδρία θα λάβει χώρα Είδαμε τον κανονισμό εισόδου-εξόδου, καθώς επίσης και τον κώδικα των συνόρων. Στις 31 Μαΐου είδαμε ε, και τις τροπολογίες ε, για, την, ε, για τον κώδικα ε, ε, Σέγγεν ε, και εκεί έχουμε την ειδική αναφορά στο ΕΙΠ και το ΣΥ για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε συνενετική λύση όσον αφορά το θέμα αυτό γιατί πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατόν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ευεργετηθούν ε, ε, με τον ίδιο τρόπο όπως οι πολίτες άλλων χωρών στο πέρασμα των συνόρων. Ένα άλλο σημείο αφορά την πρόσβαση των αρχών ε, με μέσα επιβολής του νόμου. Συζητήσαμε τις δέκα συμβιβαστικές προτάσεις που έστειλε το Συμβούλιο ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ε, το σημείο που εμείς λέμε όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία το λέμε και εμείς και, το, και η Κομισιόν, ενώ ε, το Συμβούλιο λέει όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία ενώ το Κοινοβούλιο θέλει όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Επίσης, ε, συζητούμε το θέμα της ε, διακράτησης ε, των δεδομένων, άρθρο 31, και το Κοινοβούλιο, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, δεν πρόκειται να αλλάξει θέση. Τα δύο στα τέσσερα χρόνια. Το Συμβούλιο θέλει να διατηρήσει πέντε χρόνια με κάποια αλλαγή σε σχέση με την αρχική του θέση όσον αφορά τα ειδικά βιομετρικά συστοιχεία. Επίσης συζητήσαμε για τις διμερείς ε, συμφωνίες. Εδώ ενδεχομένως θα προκύψει, θα υπάρξει μια ρήτρα ε, αναθεώρησης ε, στα πέντε χρόνια. Αλλά ακόμα και αυτό το ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, δεν έχει κλείσει, είναι ακόμα ανοιχτό. Όσον αφορά το τελευταίο σημείο το οποίο είναι ακόμα εκρεμές, αφορά την ε, άρνηση εισόδου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να διατηρήσει το θέμα των αλφαψηφιακών ε, ε, στοιχείων, ενώ το Συμβούλιο αναφέρεται σε βιομετρικά στοιχεία. Και αυτό λοιπόν παραμένει ανοιχτό και περιμένουμε ε, συμβαστικές ε, προτάσεις. Πρέπει να σας πω κύριε Πρόεδρε ότι είμαι αισιόδοξο και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε συμφωνία ε, και μάλιστα πριν ολοκληρωθεί η παρούσα Προεδρία. Ωστόσο, θα ήθελα να ζητήσω από την Γραμματεία, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, να μην ε, προγραμματίσουμε κανέναν πολιτικό ε, ε, τριμερή διάλογο στις, ούτε στις 26 ούτε στις 27 του μηνός διότι έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές δεν θέλω τώρα να πω λεπτομέρειες Αυτά ήθελα να σας πω. Εάν οι συνάδελφοι θέλουν να μου υποβάλουν ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή τους, παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ε, συναδέλφους. Ε. Σημειώσαμε τις ημερομηνίε που μας επισημάνατε. Θέλει κανένα να πάρει το λόγο. Και επίσης να δω κατά πόσο θέλει να πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Συμβουλίο, η Προεδρία. Η Προεδρία θέλει να πάρει το λόγο, να πει δύο λόγια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Δίας Νεμέρα για την παρουσίασή, σου, παρουσίασή του σήμερα. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω τη δέσμευσή του Συμβουλίου και της Προεδρίας όλος ο ιδιαίτερος να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό και εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά στο Συμβουλίο για να πετύχουμε συμφωνία και σε βιβασμό για να μπορέσουμε να βρούμε συμφωνία με το Κοινοβούλιο και να ολοκληρωθεί το θέμα αυτό μέχρι το τέλη της Προεδρίας. Να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο και τους Κιώδης για τη δουλειά και προσβλέπουμε στη μελλοντική συνεργασία προκειμένου να καταφέρουμε να βρούμε συνένεση και συμφωνία μέχρι το τέλη της Μαλταζικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κανείς να πάρει το λόγο, να ευχαριστήσω τον κύριο Στία Δεμέρα για την σκληρή δουλειά που έχει αφιερώσει στο θέμα αυτό, να έχουμε υπόψη και τι ημερομηνίε που όρισε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορούμε τώρα να περάσουμε στην κώδικα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι θεωρήσει και να ε, περιμένουμε λίγο να καθίσει ο κ. Λόπος Αγγιλάρ και να περάσουμε στην παρουσίαση του πώ έχουν εξελιχθεί οι τριμερεί διάλογοι. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε, που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και φυσικά σας ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά ήθελα να παρουσιάσω στα μέλη της Επιτροπής πώς έχουν τα πράγματα σε διαφορά του τους τριμερείς διαλόγους. Καταρχάς, ε, καλώς ορίσω αυτή την ευκαιρία γιατί πρόκειται για μια σημαντική, ε, ένα σημαντικό νομοθέτημα και καλώς ορίζω το γεγονός ότι στην σύνοδο αυτή η Επιτροπή ελπίζουμε να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί μας, γιατί θα πρέπει να έχουμε υπόψη ναι, πόσο δύσκολο είναι αυτό το θέμα και πόσο ακαθόδη θέματα α, περιλαμβάνει. Εξ αρχής το Συμβούλιο ήταν ε, α, απρόθυμο να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο. Δεν υπήρξε πνεύμα καλής συνεργασία και αυτό για κάποιους λόγους συγκεκριμένου. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση πριν από τέσσερα χρόνια για την αναθεώρηση του σχετικού νομοθετήματος. Ήταν πολύ διαφορετική η πολιτική κατάσταση από τη σημερινή προφανώ. Καταρχάς ο, ο κώδικας για τι θεωρήσεις παρουσιάστηκε ως ένα εργαλείο για την οικονομική ανταλλαγή και την ανταλλαγή αμα, εργαζομένων ω κινητήριο δύναμη για την αντιμετώπιση τη κρίση, Αλλά στη συνέχεια, στην τελική ανάλυση, ο κώδικας για τις θεωρήσεις τελικά παρεμποδίστηκε από το σενάριο της ε, λεγόμενης ε, προσφυγικής κρίσης, της ε, τρομοκρατικής απειλής και έχει καταστεί τελικά ένα θέμα το οποίο έχει επιμολυνθεί από την ιστερία που έχει ξεσπάσει για τα θέματα ασφάλειας. Δικαιολογημένα φυσικά έχουν τεθεί τα θέματα αυτά και έχουν ε, αναζωπηριωθεί μέσα από κάθε τρομοκρατική επίθεση, αλλά ο κόσμος έχει αλλάξει. Και ένα παράδειγμα είναι λοιπόν ότι το θέμα των θεωρήσεων πλέον έχει παραγωνιστεί. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες λοιπόν στο πακέτο αυτό, όλοι θα περίμεναν παραπάνω δυναμισμό και το Συμβούλιο και φυσικά από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά αυτά, όπως σας είπα, πλέον αποτελούν παρελθόν. Το θέμα λοιπόν έχει μπλοκαριστεί. Η αναθεώρηση του κώδικα για τις θεωρήσεις έχει αναχαιτιστεί και γίνονται συζητήσει για το κατά πόσο θα υπάρχουν ανθρωπιστικές θεωρήσεις ή όχι και κατά πόσο θα συμπεριληφθούν. Αλλά το Συμβούλιο ούτε μία πρόθεση έχει δείξει να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι μόνο επί του θέματο αυτού, αλλά και επί μία σειρά άλλων θεμάτων. Για εμά τώρα, ω βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το θέμα δεν είναι άσπρο-μαύρο, προφανώ. Φυσικά δεν τηρούμε στάση άτεγκτη ότι αν δεν συζητήσετε για τα θέματα ανθρωπιστική θεώρηση δεν σα μιλάμε κι εμεί. Όχι, προσπαθούμε να βρούμε ένα συμβιβασμό, να ξεμπλοκαριστεί η κατάσταση. Αλλά βλέπουμε πόσο α, πραγματικά άτεγκτο είναι το Συμβούλιο και απρόθεμο να συνεργαστεί και να κάνει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Λέει δηλαδή ότι αν το Κοινοβούλιο δεν ε, παρατηθεί όλων των τροπολογιών του, δεν θα υπήρξε οποιοδήποτε συμβιβασμό. Δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε συμβιβασμό. Άρα, με σαφήνεια σα το λέω ότι δεν μπορώ να δεχτώ να αποσύρω όλε, μα όλε τι τροπολογίε. Όχι μόνο για τι ανθρωπιστικέ θεωρήσει, αλλά και φυσικά οι ανθρωπιστικέ θεωρήσει να αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα τη περαιτέρω συζήτηση. Το επιχείρημα ότι δεν είναι εδώ το σωστό σημείο να συζητήσουμε τις ανθρωπιστικέ θεωρήσει. Μα το έχουν προβάλει πολλάκι. Ρωτούμε λοιπόν. Θα μας την διαφορετική πρόταση για τι ανθρωπιστικές θεωρήσει. Αυτό αποτελεί άλλωστε πάγιο αίτημα όλων των think tank, των ε, εκκλησιών ακόμα, ακόμα των ε, ΜΚΟ που ζητούν από το Κοινοβούλιο επανελειμμένα να δώσει μια τέτοια, να ανοίξει ένα τέτοιο δρόμο για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Το έχουμε θέσει επανελειμμένα το θέμα αυτό τα τελευταία χρόνια με την υποστήριξη των σκιωδών. Συλλαμβανομένη και του σκιώδη του ΕΛΚ, του κ. Μπέκερ. Ξέρουμε πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την πρόταση για την για την επανακατάσταση και ε, έχουμε παρουσιάσει ένα non-paper για, τον, για τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε ότι η επανακατάσταση δεν αρκεί. Γιατί είναι περιοριστικό από γεωγραφική άποψης ε, και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε κατάσταση που θα είχε εφαρμογή στο θέμα της ανθρωπιστικής θεώρησης, αλλά στην τελευταία τεχνική συνάντηση τονίστηκε ότι θα υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις για να αναπτυχθεί το θέμα περαιτέρω. Και προσφάτως είχαμε συζητήσεις ε, με τον Επιτροπό Αβραμόπουλο και με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς και επιμείναμε, επιμείναμε να υπάρχει σαφής και ρητή δέσμευση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρξει το θέμα της ανθρωπιστικής ε, θεώρησης και να συμπεριληφθεί στο θέμα της επανεγκατάστασης. Άλλη μία όμως ε, προϋπόθεση που μα θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το θέμα τη γενικής διευκόλυνσης που είναι βασικό για το θέμα των θεωρήσεων και το θέμα τη συνεργασίας για την επανεισδοχή, συνεργασία λέω για την επανεισδοχή. Αυτό θα μπορούσαμε με επικοδομητικό τρόπο να το συζητήσουμε. Θα ήμασταν αντιτεθειμένοι να καταλήξουμε σε κάποιο είδου συμβιβασμό. Πέραν τούτου, η απροθυμία του Συμβουλίου δεν περιορίζονται, όπω σα είπα, στι ανθρωπιστικέ θεωρήσει, αλλά και στι υποχρεωτικέ συστάσει και στην επανένωση των οικογενειών. Επ' αυτόν θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα blank spots, αυτά τα λευκά σημεία, τα κενά σημεία, θα πρέπει να τα φροντίσουμε. Δηλαδή, να μην υπάρχει παρουσία μιας χώρας σε πρωτεύουσα άλλης χώρας όταν τίθεται θέμα ανθρωπιστικής θεώρησης. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε σε ό,τι αφορά την ε, υποχρέωση, την υποχρεωτική εκπροσώπηση. Αυτό αποτελεί ένα εργαλείο. Σε ό,τι αφορά τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Τέλος. Βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος της Μαλτέζικης Προεδρίας και θα ήθελα παρεπιπτόντως να επενέσω ιδιαίτερω τι προσπάθειε που έχουν καταβάλει από πλευρά τη Μαλτέζικη Προεδρία οι αντιπρόσωποι. Τουλάχιστον δείχνουν μια προθυμία οι άνθρωποι να βρουν μια δικοδομητική λύση. Γιατί έχουμε δείξει και κάποιοι, έχουμε δει και κάποιες προεδρίες που δεν έχουν οποιαδήποτε διάθεση συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι το Συμβούλιο πρέπει να επιδείξει και κάποια διάθεση συνεργασίας. για να καταθέσει μία ξεχωριστή πρόταση για την ανθρωπιστική θεώρηση για τα ανθρωπιστικά ζητήματα. Η διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι δεσμευμένη και αποφασισμένη να πετύχει κάποιο αποτέλεσμα. Να πετύχει μία συμφωνία προκειμένου να ολοκληρωθεί το ζήτημα αυτό επιτέλους. Θα ήθελα να ακούσω τι έχουν να πούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Έχω τη διά, την εντύπωση ότι κάτι έχει συμβεί, κάπως έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Και ενώ παλιά ήταν ε, αρνητική η στάση, τώρα ενδεχομένως να υπάρχει κάποια διαλλακτικότητα. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τις συζητήσεις χωρίς το θέμα των ανθρωπιστικών θεωρήσεων, αλλά θα πρέπει να επιδείξουμε μια διάθεση συμβιβασμού για τα υπόλοιπα θέματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επαναλαμβάνω, μπορεί να δείξει ε, κάποια διάθεση συμβιβασμού για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις, αν δείξει κάποια διάθεση συμβιβασμού και το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά την επανένωση οικογενειών, για παράδειγμα. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά να το τονίσω αυτό. Έχουμε μια κατάσταση όπου το Συμβούλιο δεν ενδιαφέρεται να υπάρξει νομοθεσία στο θέμα της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και της ασφάλειας, εκτός και αν κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω. Σε σχέση με το τρέχον status quo. Αυτό είναι απαραδεκτό για το Κοινοβουλίο. Ναι, κοιτάξτε. Έχουμε και την επόμενη έκθεση για την ιδιωτική σφαίρα, την ιδιωτική ζωή και μετά έχουμε και τις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μονικά που εκπροσωπεί τον κύριο Μπέκερ ο κύριος Ζεράρ Ντεπρέ και μετά ολοκληρώνουμε το θέμα αυτό. Η κυρία Ολμαϊρ, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θεωρώ ότι η ανθρωπιστική κατάσταση και οι ανθρωπιστικές θεωρήσεις ε, που εκδίδονται από τη χώρα μου είναι κάτι πολύ θετικό, αλλά θεωρώ ότι αποτελεί όντως το λαθό ε, φάκελο. Αυτό εξακολουθεί να υποστηρίζει ως θέση το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το να βρούμε εδώ μια σωστή λύση δεν μπορεί να σχετίζεται με τους τουρίστες, με τους ε, εμπόρους και τις θεωρήσεις τους. Ο κύριος Μπέκερ ε, μου έδωσε σαφή εντολή και η συναδελφία από το ΕΛΚΑ ότι θα θέλαμε οι έμποροι και οι τουρίστες να έχουν μια πιο απλοποιημένη διαδικασία γιατί Νομίζω ότι είναι δύσκολο να μιλάμε για ιστερία σε ό,τι αφορά για τέτοια θέματα ασφάλειας. Διαπιστώνονται διαπιστώνονται από τα πλευρά των κρατών μελών ότι δεν λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την ασφάλεια, ανεξάρτητα τώρα με το τι γίνεται με το θέμα της ανθρωπιστικής θεωρήσης, το οποίο δεν θεωρώ ότι ε, σχετίζεται ιδιαίτερα με το θέμα αυτό. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν κράτα-μέλη τα οποία είναι σε θέση και είναι τεθειμένοι να εκδώσουν ανθρωπιστική θεώρηση και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επίσης έχει αποφανθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να επιβάλλει μια τέτοια απόφαση στα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί να ασχίσει τέτοια πίεση και να τα υποχρεώσει να εκδώσουν ανθρωπιστική θεώρηση. Και σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα εκκρεμή ζητήματα, θα ήθελα να πω εξ ονοματο του κ. Μπέικερ σε ό,τι αφορά το θέμα τη οικογένειακή επανένωση, το θέμα της θέμα όλα αυτά τα θέματα νομίζουμε ότι θα ήταν πιο εύκολη η επιτευξή συμφωνίας. Κατά πόσο θα είναι ξεχωριστή η πρόταση για την ε, ανθρωπιστική θεόραση ή κατά πόσο θα υπάρχει θα μπει στο θέμα της επανεγκατάστασης, είναι άλλο θέμα, αλλά γενικά σε ό,τι αφορά την νόμιμη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δύο υπάρχονται στο θέμα αυτό και για τους πρόσφυγες, αλλά να πιστεύουμε Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή λύση για τους εμπόρους και τους τουρίστες. Το θέμα τώρα ότι τα κρατημέλη δεν δε, να βγάλουν ε, άμεσα ε, θεωρήσεις για άτομα τα οποία δεν έχουν οποιοδήποτε ταυτότητα και βρίσκονται στα σύνορά του, πρέπει να πω ότι το καταλαβαίνω από κάπου και θεωρώ ότι θα πρέπει να επιδείξουμε ε, μια διάθεση και να είμαστε και λογικοί και χρειάζεται να βρούμε ένα νόμιμο διάδρομο για τους πρόσφυγες, το οποίο όμως θα πρέπει να ρυθμιστεί σε ξεχωριστό νομοθέτημα. Ευχαριστώ πολύ. Η Χέλγα Στίβενς είναι πρώτα από το ECR, μετά εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Καλημέρα σε όλους. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό και το πώς έχει εξελιχθεί. Ξεκίνησε μία, ως μία αναθεώρηση των ε, υφιστάμενων διατάξεων για τις θεωρήσεις και τότε προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε με πιο εύκολο και ευέλικτο και γρήγορο τρόπο το θέμα των θεωρήσεων για τους πολίτες μέσω, για παράδειγμα, μιας της σελίδας μέσω της οποίας μπορεί να γίνει το αίτημα. Το ε, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ζήτησαν να μπει το θέμα της ανθρωπιστικής ε, θεώρησης στην νομική αυτή πρόταση. Ακόμα παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αναφαντών κατά σε ό,τι αφορά τις ανθρωπιστικές ε, θεωρήσεις, σε ό,τι αφορά τη χορήγηση τέτοιων θεωρήσεων από τα προξενία άλλων χωρών. Το Κοινοβούλιο είχε αποφασίσει πέρα, αλλά από νομική άποψη δεν στέκει αυτό. Το, ελεκτικό, η, η, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε πρόσφατα, αποφάθηκε πρόσφατα, δεν είναι το να επιβάλλεται τέτοια υποχρέωση στα κράτη-μέλη. Ή το αίτημα των σοσιαλιστών και δημοκρατών, λοιπόν, τότε έπρεπε να αποσυρθεί, Όπω είχε ζητήσει και το Συμβούλιο. Δεν έγινε όμω κάτι τέτοιο και το αποτέλεσμα είναι να είναι κατά τη πρόταση αυτή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την εντύπωση ότι πολλοί σκιώδει ε, εισηγητέ είναι αντίθετοι προ την εξέλιξη των πραγμάτων. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητέ κυρία εισηγητά, σα το ζητώ επανειλημμένα. Αφαιρέστε οποιαδήποτε αναφορά σε ανθρωπιστικέ θεωρήσει και συνεχίστε τι διαπραγματεύσει, γιατί θα ήταν πραγματικά ντροπή να, μπορέσουμε, να μην μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο αυτό μέχρι το τέλη της μα. μας. Ευχαριστώ πολύ. Και τέλο ο Ζεράρ Ντεπρέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή μας. Ως σκιώδης είχα την ευκαιρία να εκτιμήσω την προσήλωσή του σε αυτό το φάκελο και το πόσο ε, θέλησε να διαβουλευθεί με όλους τους σκιώδης. Πραγματικά, ειλικρινά τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ε, τώρα, σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα, έχει δίκιο. Το Συμβούλιο δεν ανοίγει πολύ το παιχνίδι όσον αφορά την διευκόλυνση του συστήματος των θεωρήσεων. Αυτό είναι προφανές και πρέπει να συνεχίσουμε. Έγινε μια ψηφοφορία στην Επιτροπή μας, έχουμε μια εντολή, άρα πρέπει να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε αυτήν τη μας τη θέση. Δεν είμαι, όπως μόλις είπε η κυρία Στέβενς, εγώ υπέρ της ε, αλληλέγγυας ψήφου υπέρ της ε, ανθρωπιστικής θεώρησης. Αντίθετα, κάποιες φορές υπήρξε πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο που είπε ότι ναι, επιθετούμε ε, ε, ανθρωπιστική θεώρηση. Το ζητάμε. Το θέμα όμως είναι πώς, πού θα το βάλουμε. Είναι σαφές ότι δεν θα έχει τη θέση του στο κεντρικό στο νομοθέτημα για τις θεωρήσεις, γιατί το Συμβούλιο δεν το θέλει, η Κομισιόν διαφωνεί και η δικαιοσύνη είπε σε μια απόφαση ότι δεν είναι αυτός ο χώρος. Αυτό δεν εμποδίζει τίποτα τον αγώνα μας για την ανθρωπιστική θεώρηση. Έχουμε εντολή για να προσπαθήσουμε να το πετύχουμε. Έχει κλείσει αυτό το παιχνίδι. Όχι. Σε άλλη πρόταση όμως... Το Συμβούλιο έχει ήδη καταθέσει τροπολογίες για την επανεγκατάσταση και κάνει λόγο για ανθρωπιστική υποδοχή ανοίγει μια μικρή πορτίτσα. Δεν είναι μεγάλη η πόρτα, αλλά εμείς πρέπει να την, ε, ε, να την ε, μεγεθύνουμε. Και αυτό θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση η Κομισιόν. Το Συμβούλιο έχει ανοίξει μια μικρή πορτούλα. Η Κομισιόν όμως θα πρέπει να υποβάλει μια πρόταση ώστε να προσπαθήσει αυτή την πόρτα να την διευρύνει να τη διατηρήσει και να τη διευρύνει αν γίνεται. Άρα λοιπόν για τον κώδικα το θεωρήσουν και επί τη βάση τη εντολή που έχουμε λάβει και παράλληλα με όλα αυτά θα πρέπει να οθήσουμε την Κομισιόν να υποβάλει πρόταση. Γιατί άνοιξε όπω είπα την πόρτα το Συμβούλιο σε ένα άλλο φάκελο και είμαι πεπισμένο ότι εάν το θελήσουμε αυτό και πιέσουμε την Κομισιόν και μας υποβάλλει πρόταση, θα πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα και στα δυο μέτωπα. Και για τον κώδικα των θεωρήσεων και για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Και γι' αυτό και εμπιστεύομαι τον εισηγητή μας ώστε να μεταφράσει αυτό μας το αίτημα προς την Κομισιόν με εξαιρετικά ε, σταθερό και, και έντονο τρόπο γιατί ε, δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, μας πιέζει ο χρόνος ε, σήμερα και πρέπει να συζητήσουμε και για την ιδιωτικότητα, την ιδιωτική ε, σφαίρα, πριν από τις ψηφοφορίες. Χωρίς άλλη η περαιτέρω καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στην, στην σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την πρώτη παρουσίαση του, της πρότασης κανονισμού για τον ιδιωτικό χώρο και ευχαριστώ την Κομισιόν γιατί τώρα έχουμε εργαστεί πάνω σε αυτό το θέμα. και έχουμε συντάξει ένα καλό ε, σχέδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σημαντική αυτή νομοθεσία, γιατί συμπληρώνεται έτσι το πακέτο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπου έχουμε χώρο για το GDPR και θα εφαρμοστεί και αυτό ταυτόχρονα. ταυτόχρονα με το Γενικό Κανονισμό της Προστασίας Δεδομένων δηλαδή. Το έχουμε συζητήσει αυτό στις διάφορες επιτροπές και με τους εκπροσώπους του Γραφείου Προστασίας ε, Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 39 τι, ε, το τι δηλαδή σημαίνει ε, αυτό έχουμε κάνει εκτεταμένες διαβουλεύσεις έχουμε κάνει συνεδριάσεις με πάνω από 80 μπλεκόμενα μέρη είναι πολύ αντιφατικό το θέμα αν το δούμε από την πλευρά των χρηστών που επιθυμούν πολύ ψηλό επίπεδο προστασίας αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε κλάδο τον ε, επιχειρηματικό που ζη... που ρωτά ένα σωρό λεπτομέρειε για δει αν θα μπορέσει να τα εφαρμόσει όλα αυτά στην πράξη. Είμαι βέβαια ότι τώρα έχουμε μια σαφή εικόνα ε, για το, τα συμφέροντα που υπάρχουν και για τις αντιφάσεις που υπάρχουν. Τώρα το πρόβλημα της σχέσης του γενικού κανονισμού με το τότε εδώ τη ιδιωτική ζωή. Αυτό ο κανονισμό στηρίζεται στο άρθρο 8 τη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ η προστασία της ιδιωτική ζωής ε, βασίζεται στο άρθρο 7. Προστασία τη ιδιωτική ζωή, όχι μόνο τα στοιχεία δηλαδή τα ιδιωτικά, αλλά και οι ιδιωτικέ επικοινωνίε θα πρέπει να προστατεύονται. Και αυτά όλα βέβαια είχαν συνταχθεί όταν δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα, εφή τηλέφωνα και κοινωνικά, μέσα κοινωνικής δικτύωσης γιατί τώρα έχουμε ένα σωρό μηνύματα που πάνε και από το Messenger και ένα σωρό ε, άλλα μέσα. Και αυτό, γι' αυτό είναι τόσο σημαντικά αυτά που συζητάμε για τους χρήστες. Οι χρήστες περιμένουν να κάνουμε πολύ καλή δουλειά ώστε να εξασφαλίσουμε ψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής οι ανησυχίες είναι πολλές, όπως δείχνουν οι έρευνες, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και στην ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε πως είναι κανονισμός, να είναι κανονισμός γιατί είναι σαφές εφόσον υπάρχει ενιαία αγορά ότι οι κανόνες θα πρέπει να είναι οι ίδιοι για όλους. Ωστόσο, ε, τα κράτη-μέλη έχουν την κυριαρχία όσον αφορά την προστασία ε, των δεδομένων. Ε, πολύ σημαντικό έργο της Επιτροπής μας θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι διατάξεις σε αυτή την νομοθεσία θα είναι σύμμορφες προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των δεδομένων, γιατί αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται αυτός και, γίνε, και ο κόσμος ε, απορεί πώς όλα αυτά θα συνδυαστούν. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ευθυγράμμιση του νομοθετήματος αυτού, δεν μην δοθεί νέα ερμηνεία σε κανένα από αυτά τα άρθρα. Πρέπει επίσης να προστατεύσουμε την ιδιωτική ζωή όχι μόνο στη μετα γραφή ας πούμε στοιχείων αλλά και όταν, όσον αφορά τους ίδιους ε, τις συσκευές ε, των χρηστών γιατί ξέρουμε ότι τα εφηή e μας τηλέφωνα ακόμα και οι τηλεοράσεις μας ε, έχουν τεράστιες δυνατότητες αποθήκευσης πληροφοριών γι' αυτό πρέπει και αυτό το ζήτημα να το χειριστούμε όπως και στο γενικό κανονισμό στόχος μας είναι να έχουμε να δώσουμε έμφαση στις, ε, στην προστασία, αλλά ταυτόχρονα να βάσει αυτού του κανονισμού είναι η συγκατάθεση η προσωπική. Να αναγνωρίζουμε βέβαια τα θεμητά ενδιαφέροντα και συμφέροντα του κλάδου, αλλά όταν πρόκειται για ιδιωτική συνδιαλλαγή θα πρέπει ε, να ε, δίνει τη συγκατάθεσή του και ο εκάστοτε ιδιώτης για τη χρήση των δεδομένων του. Τώρα, παράδειγμα, άρθρο 39 πολύ καλές συμβουλές για το πώς θα βρεθούν καλύτερες λύσεις. Οπότε τώρα αρχίζουμε να εργαζόμαστε πάνω στις λεπτοφέρειες. Σε δύο εβδομάδες, 21 Ιουνίου μάλιστα, σκοπεύουμε να υποβάλουμε την πλήρη έκθεση ώστε να γίνει πλήρη συζήτηση στην Επιτροπή για να λάβουμε τις τροπολογίες σας πριν τις ε, θερινές διακοπές και να επιστρέψουμε από τις θερινές διακοπές με έτοιμο κείμενο ώστε να ξεκινήσουμε την επεξεργασία του με τους σκιώδεις από τις αρχές Σεπτεμβρίου για να διατηρήσουμε αυτές τις ε, κατευθύνες γραμμές. Επίσης, η Εστονική Προεδρία αναμένεται να εργαστεί εντατικά για το θέμα αυτό και για την ε, νέα ψηφιακή αγορά. Να ευχαριστήσω τους Κιώδης που έχουν περιλάβει, που έχουν ε, μάλλον ε, ε, συμμετέχει σε αυτήν την παρασκευαστική εργασία. Έχουμε ήδη με τον κύριο Μπόνη προετοιμάσουμε τέσσερα σεμινάρια. Πολύ εντατικές ημερίδες, αλλά έτσι μπορέσαμε να καταλάβουμε τι διακυβεύεται. Ευχαριστώ λοιπόν. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Το περιμέναμε πολύ καιρό το θέμα αυτό να συζητηθεί. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που έχουμε τώρα και την πρώτη εντελεγή ε, απόψεων. Δεν έχουμε δυστυχώς πάρα πολύ χρόνο ε, σήμερα το πρωί, αλλά νομίζω ότι αν χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο σωστά θα καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Ο κύριος Αμπόνη, η κυρία Στίβενς, ο κύριος Αλμπρέκτ. Ιντβελτ, ε, δεν ξέρω αν θέλει και κάποιος άλλος να πάρει το λόγο, γιατί θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Ωραία, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να τα κάνουμε όλα έγκαιρα. Κύριε Μπόνι, παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Ε, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να πω ότι ευχαριστούμε την Κομισιόνα ε, γιατί παρουσίασε το θέμα αυτό. Θα ήθελα βέβαια ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια όχι μόνο για τα σημερινά τη σχόλια αλλά ε, και για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε και με τον οποίο ηγήθηκε των τεσσάρων αν δεν κάνω λάθος των τραπεζών που κάναμε μέχρι τώρα ε, συζητώντας ε, για τον κανονισμό αυτό ε, συζητήσεις οι οποίες έδειξαν ότι χρειαζόμαστε τη μορφή του κανονισμού για αυτό το νομοθέτημα και για τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία εκκρεμούν ακόμα να βρούμε κάποια λύση. Ας πούμε την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων με βάση των νέων στοιχείων και βεβαίως και σε σχέση και με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Βεβαίω, τα ζητήματα της ασφάλειας ε, των επικοινωνιών και το θέμα τα απορρίτου των επικοινωνιών είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να δούμε πώς θα τα διασφαλίσουμε και επίσης ε, πώ ε, θα καλύψουμε τους τελικούς χρήστες και τα τερματικά τα οποία βρίσκονται στα σπίτια, πώς θα τα προστατέψουμε και αυτά. Ε, και όλα αυτά βεβαίως ε, προφανώς ε, με σεβασμό των όσων αναφέρονται στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων γιατί αυτό που θέλουμε είναι να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων όχι να τους δημιουργήσουμε επιπλέον προβλήματα Παρακολουθεί, βεβαίως εξακολουθεί να υπάρχει και το θέμα του χρόνου θέση σε ισχύς του κανονισμού ταυτόχρονα δηλαδή με τον ΓΚΠΔΕΛΤΑ. Και το ερώτημα είναι εάν θα μπορέσουμε και από τεχνικής απόψεως να έχουμε πλήρη υλοποίηση. Από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί εν τέλει το άρθρο 11 γιατί ιδιαίτερος προβληματίζομαι εγώ γιατί δεν είναι σαφής η δυνατότητα των κρατών μελών να αλλάξουν ή όχι και υπάρχει η δυνατότητα ε, ε, να προκύψει σενάριο το οποίο θα καταστρέψει πλήρως ε, τις όσες προσπάθειες έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα. Από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε ποιες θα μπορούσαν να είναι οι απρόσμενες ή απρόβλεπτες επιδράσεις ή ο απρόβλεπτος αντίκτυπος αυτών των διατάξεων κυρίως επί των επιχειρήσεων. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να ε, ε, καταλάβουμε ε, ακριβώς περί τίνος πρόκειται και ποια είναι η πρόκληση όσον αφορά τον κανονισμό αυτό, τι σημαίνει δηλαδή η συνεργασία με τους εταίρους, να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι εταίροι και βεβαίως να δώσουμε και την δυνατότητα ενεργούς ελεύθερης επιλογής των τελικών χρηστών χωρίς να λησμονήσουμε όμως και κάποιες, ε, κάποια κίνητρα που θα πρέπει να δώσουμε στις επιχειρήσεις έτσι ώστε να βελτιώσουν ε, την ε, ασφάλεια και το απόρριτο. Αυτά μέχρι τώρα και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για, τους πολύ για τις πολύ χρήσιμες τρογγυλές τράπεζες που οργάνωσε. Κυρία Χέλγκα Στίβενς. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ μιλάω εξ ονόματος ε, του σκιώδου συζητητού της ομάδας μου που δυστυχώς, Αντόλτον, ε, που δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι παρόν. Ε, άποψή του είναι ότι ε, με σκεπτικισμό βλέπουμε ακόμα την πρόταση αυτή έχουμε κάποιους προβληματισμούς ε, γιατί θα πρέπει ε, μέχρι το Μάιο του 2018 να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες και να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός μαζί με το Γενικό ε, Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα αντιμετωπίσουν το άχθος αυτό οι επιχειρήσεις οι οποίες ταυτόχρονα θα πρέπει να υλοποιήσουν, να εφαρμόσουν και τους δύο κανονισμούς. Με το προσαρμοσμένο Γενικό Κανονισμό ε, ήδη οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προετοιμαστούν ε, για την θέση ισχύ του κανονισμού αυτού. Ο εισηγητή ε, του ECR θεωρεί ότι θα πρέπει πρώτα να ε, υλοποιηθεί, να εφαρμοστεί μάλλον ο γενικός κανονισμός, να δούμε τα ενδεχόμενα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν και μετά να ισχύσει ο άλλος κανονισμός. Γιατί αυτός ο δεύτερο κανονισμός ενδεχομένως θα έχει κάποιον απρόσμενο αντίκτυπο, κυρίω σε νεοφυείς επιχειρήσεις, startups. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει ε, να δούμε τις, ε, τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει μέχρι τώρα γιατί έχουμε και στο διαδίκτυο και στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες έχουμε προβλήματα όσον αφορά ριζοσπαστικοποίηση κλπ. Μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να τα ξεπεράσουμε. Επίσης το ίντερνετ των πραγμάτων θα πρέπει να μας απασχολήσει. Επίσης, ε, οι επιχειρήσεις πολύ ε, απασχολούνται όσον αφορά και προβληματίζονται με αυτούς τους κανόνες που αφορούν τα cookies και το tracking, την παρακολούθηση ε, των επιλογών. Πιστεύουμε ότι εδώ θα δυσκολευτούν οι επιχειρήσεις με άλλους τρόπους να προσεγγίσουν το κοινό στόχο ε, στο, το οποίο θέλουν να προσεγγίσουν. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει ε, να ε, δείξουμε μεγάλη προσοχή στα θέματα αυτά. Ε, επίσης ε, ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει πολλαπλή νομική βάση όσον αφορά τα cookies και το tracking που θα, προστατεύει όμως και τα θεμητά δικαιώματα και των χρηστών και των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Σόφι Ιντβελτ, ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ μάλιστα την εισηγήτρια για την πολύ εμπεριστατωμένη της ε, προσέγγιση, προσέγγιση ενός ιδιαίτερου περιπλόκου θέματος. Θέμα λοιπόν επί του οποίου θα πρέπει να υπάρξει σωστή ανάλυση και πλήρης κατανόηση των ε, στοιχείων έτσι ώστε αφενός να μην υπάρχουν επικαλύψεις με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων αλλά ταυτόχρονα και να αποφευθούν κενά ε, υπάρχουν αυτοί που λένε ότι δεν θέλουμε καθόλου δεύτερο κανονισμό γιατί όλα είναι μια χαρά. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό βέβαια. Πιστεύω ότι όντω υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει περαιτέρω να διευθετηθούν αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με μεγάλη σαφήνεια ε, κυρίω όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή. Δεύτερη παρατήρηση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταστήσουμε απολύτως σαφές ε, το, το ποια είναι η οικονομική αξία των δεδομένων. Μιλάμε για προστασία ε, καταναλωτών, προστασία πολιτών κτλ. Μιλάμε όμως και για καινοτομία και για ανάπτυξη. Ε, αλλά σπανίως συζητούμε το γεγονός ότι τα προσωπικά δεδομένα έχουν κοινωνική αξία, έχουν συγγνώμη, οικονομική αξία, έχουν οικονομικό βάρος πληρώνουν άνθρωποι για να πάρουν αυτά τα προσωπικά στοιχεία. Νομίζω ότι αυτό το λησμονούμε συχνά και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας σε αυτόν τον κανονισμό και να συμπεριληφθεί στον αντίκτυπο που μπορεί ενδεχομένως να έχει ο κανονισμός αυτός. Τελευταία μου παρατήρηση. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες ε, πληροφορίες σχετικά με ε, περιοχές ε, οι οποίες, ε, των οποίων μάλλον την εξέλιξη δύσκολα μπορούμε να προβλέψουμε. Ε, είναι δύσκολο να ρυθμίσει κανείς το tracking και το monitoring ας πούμε των ανθρώπων ή το, του πλήθους σε ένα ανοιχτό χώρο. Κάπως έτσι είναι και η προσπάθεια ελέγχου του tracking στο ίντερνετ και δεν μπορεί βεβαίως να λυθεί το ζήτημα μέσω του αιτήματο συνένεσης του χρήστη όσον αφορά τη συνένεση μάλιστα, όπως και η συγγήτρια και ε, ο σκιώδης ε, του ΕΛΚ, πιστεύω ε, ότι ότι η συνένεση αποτελεί πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, στοιχείο. Ξέρω ότι δεν ε, είναι πολύ άνετες ορισμένες επιχειρήσεις με το θέμα αυτό, αλλά ε, εάν το επιχειρηματικό μοντέλο μιας εταιρείας, το business model μιας εταιρείας βασίζεται στο κάνω κάποια πράγματα τα οποία θα φέρουν σε αμήχανη θέση ή θα δημιουργήσουν πρόβλημα στους καταναλωτές, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρήσουν το μοντέλο τους. Πιστεύω και ελπίζω ε, ότι τελικά θα προκύψει ένας ε, κανονισμός ε, ο οποίος θα μπορέσει να ικανοποιήσει, ίσως όχι όλους, αλλά τουλάχιστον τον μέγιστο δυνατό αριθμό εμπλεκομένων. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, first of all, also... Uh, ευχαριστώ πολύ και εγώ θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εισηγήτρια για την προπαρασκευαστική εργασία αλλά και για την καλή συνεργασία με τους σκιώδες, ιδιαίτερα τον κύριο ε, Μπόνι όπου συνδιοργανώσατε αυτές τις αρχικές συνεδριάσεις που ήταν πολύ, πολύ βοηθητικές για μας. Να στηρίξω την εισηγήτρια γιατί προσπαθεί να είναι ε, όσο μπορεί πιο κοντά στο χρονοδιάγραμμα. Γιατί βέβαια στο τέλος θα πρέπει να δούμε όλοι πού βρισκόμαστε και κατά πόσο όλα αυτά θα μπορέσουμε να τα κάνουμε και στην πράξη. Αλλά καταρχάς θα πρέπει να, να γνωρίζουμε, να περάσουμε το νομοθέτημα αυτό πριν να αρχίσει να ισχύει ο γενικός κανονισμός. Διαφορετικά θα αρχίσει να εφαρμόζεται και δεν θα έχουμε τίποτα για τον τομέα της ιδιωτικής ζωής. Τώρα, ο κανονισμός αυτός για την ιδιωτική ζωή δεν είναι τίποτα το νέο που προστίθεται στο γενικό κανονισμό, αλλά που θα είναι κάτι που θα μείνει ακόμα και αν δεν περάσει ο κανονισμός. Είναι κάτι το οποίο ρυθμίζει, είναι ειδικό τομέα, πρόκειται για την ιδιωτική ζωή, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ο λόγος για την αντικατάσταση αυτού είναι παρόμοιος με αυτόν που Λέμε ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα μόνο μέσο και μία μόνο νομική, ένα, μία μόνο, ε, ένα μόνο νομοθέτημα για κάθε θέμα παρά να έχουμε 10-15 ε, νομοθεσίες που πρέπει να μεταγραφούν στα κράτη-μέλη και βεβαίως θέλουμε να εισάγουμε και τις, τους ίδιους μηχανισμούς ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εποπτεία και την αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, Άρα λοιπόν δεν υπάρχει μόνο το δικαίωμα για την προστασία των δεδομένων, αλλά και για την μυστικότητα ή τον απόρριτο χαρακτήρα των πληροφοριών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα, αλλά και αύριο μεθαύριο που θα ασχοληθούμε το ίντερνετ των πραγμάτων. Εγώ θα ήθελα να πω πως δεν πιστεύω πως κανείς έξω θα δεχτεί κανονισμό ε, προστασίας ιδιωτικής ζωής που έχει πιο αδύναμο χαρακτήρα από τον, την ισχύουσα οδηγία για την ιδιωτική ζωή. Πρέπει λοιπόν αυτό να το, κάνουμε, να το καταστήσουμε σαφές. Πάντως ε, το χαμηλότερο επίπεδο είναι αυτό που υπάρχει τώρα στην, στην ε, οδηγία για την ιδιωτική ζωή και το συζητήσαμε αυτό πώς καταστεί τεχνικώς πιο εφικτό να έχουμε επικοινωνία ανάμεσα στο υποκείμενο των στοιχείων και τον ελεκτή των στοιχείων και το πώς αυτοί οι κανόνες θα εφαρμοστούν καλύτερα σε ιδιαίτερα όσον αφορά τις, ε, τις υπηρεσίες over the top, online, offline, με το Wi-Fi, το Bluetooth κτλ. κτλ. Δεν μπορώ. Δεν νομίζω πως θα μπορέσουμε λοιπόν να κατεβούμε κάτω από αυτό το επίπεδο. Εάν δουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει το tracking που γίνεται παντού σε κάθε διαδικασία επικοινωνία και ότι χρειάζεται περισσότερο έλεγχο και όχι λιγότερο στην πράξη. Ευχαριστώ. Ναι, λέει ο πρόεδρο, Ε, μας παρουσίασε ε, γιατί χρειαζόμαστε την οδηγία από πρακτική άποψη. Μαρίντ, η Επιτροπή θέλει νομίζω. Ένα λεπτό μπορείτε παρακαλώ. Σε ένα λεπτό να μας πείτε τι θέλετε. Και μετά θα δώσω το λόγο στη Μαρίντη για, το τελευταίο, για να κλείσει το θέμα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ουσιαστική συζήτηση. Uh, for attention you are uh, giving to this file. Uh, I αποδίδουμε μεγάλη προσοχή σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις για να βοηθήσω στη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα για αυτό το θέμα της ε, ταχεία. Ε, η μέθοδος που έχουμε ακολουθήσει για αυτή την πρόταση δεν διαφέρει από τις άλλες. Ε, ε, πρόκειται για αναθεώρηση ενό υφιστάμενου νομικού μέσου, άρα λοιπόν και μπορούμε να το εγκρίνουμε μέσα στις προθεσμίες που έχετε θεσπίσει και πιστεύω πως είναι πολύ καλό αυτό. Υπάρχει και συγχρονισμός με τις άλλες επιτροπές και την επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή όσον αφορά τις τροπολογίες αλλά και ε, οι προεδρίες θα θελήσουν να ασχοληθούν και να ολοκληρώσουν. Θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε τους νομοθέτες να προχωρήσουμε. μόνος μας στόχος είναι να πάμε γρήγορα, αλλά να, πάμε, ε, να προχωρήσουμε με ουσιαστικό τρόπο ε, με, ζει με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Στοιχείων προς όφελος των επιχειρήσεων γιατί, κυρίως γιατί θα πρέπει να το δεχτούμε ότι τα ίδια τμήματα ασχολούνται με την νομική βεβαιότητα και με την ε, προσέγγιση του συνεισηγητή μέχρι το Μάιο του 2018. Αυτό προς χάρη βεβαιότητας στην αγορά και προς χάρη ε, των χρηστών. Τώρα υπάρχουν πολύ καλά επιχειρηματικά μοντέλα στην αγορά για τα όσα περιέχονται στην πρόταση, αλλά υπάρχουν και επιχειρηματικά μοντέλα που αποτρέπουν στους χρήστες να χρησιμοποιούν καλύτερα τα στοιχεία. Άρα λοιπόν στόχος είναι μια διαφορετική αγορά Παρακαλώ, ολοκληρώστε, λέει ο Πρόεδρο. Μάλιστα, θέλουμε να βοηθήσουμε και με τεχνική αρρωγή το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Ξέρουμε πω κάνετε πολλέ συνεδριάσει και αυτό μα βοηθά πολύ και είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στην εργασία σα. Μάρια, να κλείσουμε το θέμα. Ναι, να ευχαριστήσω όλους ε, και τους κοιόδης που έχουν ήδη αρχίσει τη συνεργασία και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Επιτροπή που ήταν πολύ βοηθητική και πολύ ανοιχτή στη συζήτηση και ελπίζω πως θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ Μαρή. Εξαιρετική συζήτηση. Και το σχέδιο έκθεσης θα παρουσιαστεί στις 21 Ιουνίου. Παρακαλώ συνάδελφοι να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Είναι 10 παρά 1 λεπτό. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σε 1 λεπτό. Colleagues, if you take your seats, we'll begin the So we have Η, πρώτη ψηφοφορία λοιπόν είναι του κυρίου Πίτερσεν για την έκθεση δηλαδή του κυρίου Πίτερσεν και θα ξεκινήσουμε. Ε, αφορά τον Φορέα Ευρωπαϊκών Εθνικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Αν όλοι έχετε τις κάρτες σας και είστε ψυχολογικά έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τροπολογία 35, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Α, δεν έχουν ετοιμαστεί όλοι. Πρέπει λίγο χρόνο να τους δώσω. Monica, do you want to move? Yeah. it's a couple of colleagues who have got faulty machines. So just be patient. Εάν κάποιος ε, δει ότι δεν λειτουργεί το μηχάνημά του να μετακινηθεί. Okay, the vote is closed. Um, that's, that is... Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 14 υπέρ. Α, άρχεται μάλλον η ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρας. Carried. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Ε, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Άρχεται. Τροπολογία 16 και 37 άρχεται. Εγκρίνεται. 17 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεκα, 19 ε, εγκρίνεται. 20 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβίβασμός 2 άρχεται. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 24. Άρχεται. Εγκρίνεται. 42. Πέρας. Καταπίπτει. Απορρίπτεται. 26. Όχι, το 25. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 27. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 28. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 29 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 31 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 των ιδεολογικών σκέψεων. Πέρας. Εγκρίνεται τροπολογία 2. Πέρας. Εγκρίνεται 3. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 4. Πέρας της πληροφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Πέρας. Εγκρίνεται. 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 7. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 8. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 11. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 και 24. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 13. Ε, Πέρας. Εγκρίνεται. Διανομαστικής κλήσεως η τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 38 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Πέτερσεν. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, ε, πάλι του κυρίου Πέτερσεν. Τροπολογία 40, άρχεται η ψηφοφορία. 40, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας εγκρίνεται 14 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 41 πέρας απερίφθη τροπολογία 15 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Πέρας. Εγκρίνεται. 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 18 και 42 οι τροπολογίες, άρχεται η ψηφοφορία, επί των τροπολογιών 1842 πέρας εγκρίνονται τροπολογία 19 άρχεται πέρας εγκρίνεται τροπολογία 20 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 21 άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Εγκρίνεται. 43. Πέρας. Εγκρίνεται. 44. Πέρας. Εγκρίνεται. 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Πέρας και εγκρίνεται. 47. Πέρας. Εγκρίνεται. 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 49 πέρας εγκρίνεται. 50 πέρας εγκρίνεται. 51 πέρας εγκρίνεται. 52 πέρας απερίφθη τροπολογίες 23 και 53 από κοινού άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται τροπολογία 54 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται Τροπολογία 55. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 56. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται τροπολογία 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται τροπολογία 24. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογίες 25 και 61 από κοινού, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 26, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Αιτιολογικές σκέψεις, τροπολογία 27, άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται τροπολογία 1 πέρας εγκρίνεται τροπολογία 2 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται τροπολογίες 3 και 28 από κοινού Πέρας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 29. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογίες 4 και 30 από κοινού αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Τροπολογία 6 και 32 από κοινού άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 7. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 36. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία διανομαστικής κλίσεως επί του συνόλου του τροποποιηθέντος κειμένου. Α, πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 26 ψήφοι υπέρ, 14 ψήφοι κατά, μία αποχή. Περιμένετε λίγο μέχρι να περάσουμε στην επόμενη κατάλογο ψηφοφορία, παρακαλώ. And this is a single vote. Μία μόνη ψηφοφορία με τον κύριο Μπόνη, συγγετή για τον κανονισμό για την ανταλλαγή συστήματων έγκυρης προειδοποίησης για την αξιολόγηση κινδύνων σε ό,τι αφορά τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες. Μία και μόνη ψηφοφορία. Έναρξη παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται 39 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Συγχαρητήρια στην κύριο Μπόνη. Και φυσικά αυτό αποτελεί τμήμα ενός πακέτου. Το επόμενο θέμα με τον επόμενο ε, εισηγητή, την κυρία Χιμένες Μπεσερίλ Μπάριο. Ίδιο θέμα, αλλά ε, λίγο διαφορετικό, ελάχιστε διατάξει σχετικά με τα στοιχεία τη αντικειμενική υπόσταση των εγκλημάτων και τι ποινέ που ισχύουν στον τομέα τη παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Όσον αφορά τον ορισμό των ναρκωτικών. Και πάλι λοιπόν το κείμενο μετά από διαθεσμικέ ε, ε, διαπραγματεύσει, ονομαστική κλίση. Πέρας. Εγκρίνονται 39 ψήφοι υπέρ μία αποχή. Συγχαρητήρια στην Τρέζα, η οποία δεν είναι όμως παρούσα. Τελική ψηφοφορία. Um, Θα πρέπει κάτι να σας διαβάσω που είναι και πολύ βαρετό. Σας παρακαλώ υπομονή ζητώ. Πρέπει να σου το διαβάσω όλα. Μία τελική ψηφοφορία για την ομνημονία συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την διαχείριση μεγάλων συστήματων IT στον τομέα της ε, ασφάλειας και της δικαιοσύνης σε τη Eurojust. Πρέπει να σας διαβάσω όλα αυτά το Συμβούλιο αποφάσισε στις 19 Απριλίου να διαβουλευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια απόφαση τη Eurojust για να μνημόνιο συμφωνίες μεταξύ του Αιγιολίσα και τη Eurojust. Η εφαρμοστική απόφαση αποτελεί μέτρο το οποίο ορίζεται από το κεκτημένο βάσει του άρθρου 6 τη συνθήκη. και σύμφωνα με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το Συμβούλιο μέσα έδωσε τρει μήνε για να γνωμοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Δεδομένη τη σύντομη προθεσμία για την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ασυντονιστέ αποφάσισαν να εγκρίνουν το μνημόνιο μα τη απλοποιημένη διαδικασία. Προτείνουμε λοιπόν να εγκρίνουμε το σχέδιο εφαρμοστική απόφαση του Συμβουλίου με απλοποιημένη απόφαση χωρί τροπολογία βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού. Υπάρχουν αντιρρήσει, παρακαλώ. Έβγαλα και πολύ κείμενο. Γιατί δεν θέλω να σας ε, κάνω να βρεθείτε με διαβάζω για 10 λεπτά κείμενο. Αντιρρήσει. Όχι, δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Μάλιστα. Α περάσουμε στην ψηφοφορία λοιπόν. Έναρξη ψηφοφορία. Περάσει. Εγκρίνεται 37 ψήφι, μία κατά και μία αποχή. Σας ευχαριστούμε Τόμα, σας ευχαριστούμε Τόμας, πραγματικά είμαστε ανακουφισμένοι. Σας ευχαριστώ και ολοκληρώθηκαν έτσι οι ψηφοφορίες αγαπητοί συνάδελφοι. We will just pause. We have a... Να κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί έχουμε στις 10.30 ένα θέμα το οποίο είναι το 12 τη ημερήσια διαταξή και το 13 από κοινού κοινή συζήτηση με τον Ιταλό, ο Υπουργό. Αν θα μπορούσατε παρακαλώ να εξέλθετε ησύχως από την αίθουσα, αν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε. Σας ευχαριστώ.

Uh, συνάδελφοι, να ετοιμαστούμε για να εξετάσουμε το επόμενο μας σημείο. Είναι το σημείο 12 και 13 ε, στην ημερήσια διάταξη. Θέλω να καλωσορίσω τον Ντομένικο Μαντσιόνε, που είναι υφυπουργό του Υπουργείου Εσωτερικών της Ιταλίας, υφυπουργός εσωτερικών δηλαδή της Ιταλίας, ε, Σημείο που συνδυάζεται με τη σημαντική αποστολή τη Επιτροπή Λίμπε στην Ιταλία με αντικείμενο τη μετανάστευση και το άσυλο και έλαβε χώρα 18 με 21 Απριλίου. Αυτή η αντιπροσωπεία, τη οποία ηγείται ο συμπρόεδρο ή συμπρόεδρο αυτή τη Επιτροπή, η Ντίσκα και ο Χωάντα Φερνάντο Λόπε Αγγιγιάρ που θα έρθει σε λίγο. Επισκεφθήκαμε την Ιταλία λοιπόν από τι 18 στι 21 Απριλίου με στόχο να βρούμε στοιχεία και να διερευνήσουμε την κατάσταση που επικρατεί επιτόπου σε σχέση με την εφαρμογή του ε, πολιτικής ε, ασύλου και μετανάστευσης, καθώς και για να ενημερωθούμε για την κατάσταση και την πρόοδο, ε, να δούμε δηλαδή με τα ίδια μας τα μάτια τι συμβαίνει. Είχαμε επισκεφθεί καταβλισμούς υποδοχής και σημεία απόβασης, αποβίβασης μάλλον, καθώς και το, το hotspot Στη διάρκεια της αποστολής, εκπρόσωποι των τελικών αρχών, διεθνών σωμάτων, ενώσεων ε, του UNHCR, της είπα της αρμοστίας του για τις πρόσφυγες, αλλά ε, και πολλοί άλλοι ήρθαν σε μαζί μας, αλλά θα αφήσω τον συνάδελφο Υπουργό να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Καταλήξαμε σε, σε συμπεράσματα και συστάσεις που θεωρούμε πως ήταν σημαντικό να τα συζητήσουμε και γι' αυτό είμαστε πολύ ευτυχεί που είστε σήμερα εδώ. Είναι ορισμένοι εδώ από τα μέλη εκείνης της απαστολής. Σα ζητήσω λοιπόν να καταρχά να μα παρουσιάσετε τι δικέ σα απόψει, ίσω κάπω σύντομα, γιατί ίσω είναι καλύτερο να ε, ε, έχουμε περισσότερο χρόνο για συζήτηση με του συναδέλφου για τα όσα είδαμε εκεί και να μπορέσουμε έτσι να συζητήσουμε. να σας παρουσιάσουμε πώς έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα hot spots και να μας πείτε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην Ιταλία στην παρούσα φάση και μετά να ξεκινήσουμε μια συζήτηση και όπως βλέπετε έρχονται όλο και πιο πολλοί βουλευτέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας λοιπόν σήμερα και είσαστε πραγματικά ευπρόσδεκτοι εδώ. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πρέπει να πω ότι είμαι ιδιαίτερο ευτυχής ε, που βρίσκομαι εδώ σήμερα μεταξύ σας έτσι ώστε να συζητήσουμε το ε, θέμα αυτό που είναι φλέγον. Πρέπει να πω ότι η Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ επισκέφθηκε την Ιταλία πρόσφατα και ήδη είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ε, μία σειρά ε, θεμάτων που άπτονται ακριβώς ε, του ζητήματος που μας απασχολεί. Τρία είναι τα ειδικότερα, σημαντικότερα ζητήματα για μας. Το πρώτο είναι ε, τη πολιτική των hot spots ε, που η Επιτροπή είδε επιτόπου και επί του πεδίου της δράσεως, διότι ε, γιατί είχαν την ευκαιρία τα μέλη της Επιτροπής να επισκεφτούν το Ποτσάλο, αλλά έχουμε και άλλα τα οποία λειτουργούν και κάποια hot spots τα οποία τώρα δημιουργούνται. Ε, η, ιδέα των hot spots δεν είναι σαφώς καθορισμένη ε, βάσει του ε, κανονισμού και πρέπει να πω ότι όσον αφορά τα hot spot πάντα η ιταλική αντιμετώπιση βάσει της οικίας νομοθεσίας είναι πολύ συγκεκριμένη. Εμείς μιλάμε για κέντρα τα οποία δεν είναι πολύ διαφορετικά από τα άλλα κέντρα υποδοχής τα οποία είχαμε στην επικράτειά μας και κυρίως κυρίως ε, δε ε, στα νησιά ε, και στην Σικελία ιδιαίτερως αλλά και στην Καλαβρία, στις Πούλιες και στην Καμπανία. Βρίσκονται εκεί αυτά τα hot spots, αυτοί οι καταβλισμοί διότι η μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών φτάνουν ακριβώς από την Μεσόγειο και ο ασφαλέστερος ασφαλής, ο, ο, ασφαλής ε, λιμένας ε, είναι αυτός ο οποίος καθορίζεται έτσι ώστε να αποτελεί σημείο πρόσδεσης όλων των ε, πλοίων ε, Ιταλικών και άλλων είτε πρόκειται δε για πλοία εμπορικά που υποβοηθούν το έργο είτε πρόκειται για στρατιωτικά είναι σαν τα κανονικά ε, κέντρα, εντός των οποίων όμως υπάρχει υποχρεωτική ταυτοποίηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, δεν είναι ε, δυνατόν να κρατηθούν τα άτομα αυτά ε, για μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα και επομένως η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη και οπωσδήποτε και οι δικαστικές αρχές παρεμβαίνουν σε περίπτωση που ξεπεραστεί αυτό το χρονικό περιθώριο. Μέσω των μηχανισμών που έχουμε εμείς εφαρμόσει και στους οποίους έχουμε δώσει και κάποια ευελιξία ε, μέσω ας πούμε και κινητών μονάδων hot spots ε, οι αρχές της Ιταλίας έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν όλα τα άτομα τα οποία έχουν αποβιβαστεί στην Ιταλική επικράτεια. Πρόκειται για μια επιχείρηση την οποία εγώ θεωρώ η οποία εγώ θεωρώ ότι παρόλα παρόλα τα προβλήματα που έχουν ε, παρουσιαστεί, τη θεωρώ έλεγα ε, σημαντική και χρήσιμη. Πρώτον ε, και κυρίως διότι κανένας μηχανισμός και καμία δομή υποδοχής, κανένα σύστημα υποδοχής δεν μπορεί να οργανωθεί, όχι μόνο στη χώρα μου αλλά και σε όλη την Ευρώπη, εάν δεν γνωρίζουμε πόσα και ποια άτομα φτάνουν στην επικράτειά μας. Το δεύτερο στοιχείο, η δεύτερη κύρια αιτία είναι ότι όλο και συχνότερα διαπιστώνουμε ότι η υποδοχή θα πρέπει να έχει παράλληλα και ένα σύστημα ασφάλειας. Ε, ε, πράγμα βεβαίως και διαπίστωση η οποία έχει επιδράσει ε, σε μία σειρά αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κάποιες αποφάσεις όπως ας πούμε αυτή της επανεισδοχής οι οποίες αποφάσεις έχουν δημιουργήσει σε μερικές περιπτώσεις ακόμα περισσότερα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει όμως, ε, ε, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο να μην ξέρουμε ποια άτομα αφορά το relocation. Στην ε, χώρα μας πάντως χρησιμοποιήσαμε πλήρως όλες τις αποφάσεις και όλα τα μέσα γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως έχουμε ταυτοποιήσει όλους όσοι έχουν αποβιβαστεί στην επικράτειά μας και γνωρίζετε ότι οι αριθμοί είναι μεγάλοι. Πέρσι και ε, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι η διαδρομή της Μεσογείου είναι αυτή που οι περισσότεροι μετανάστες έχουν ε, έχουν επιλέξει είτε ε, ερχόμενοι από την Αφρική είτε ερχόμενοι και από την Ανατολή οι αφήξεις ξεπέρασαν τις 181.000. Επομένως και μετά από την ε, συνεργασία και την ε, ακρόαση ορισμένων ε, δικαστικών εκπροσώπων και σε συνεργασία και διαβούλευση με κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες πραγματικά παρουσίασαν το έργο τους στην Επιτροπή Άμυνας του Εθνικού μας Κοινοβουλίου και διαπιστώσαμε τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται διαπιστώσαμε λέω ότι το πλαίσιο είναι τόσο περίπλοκο και ότι ε, είναι τόσο διαφορετικές οι καταστάσεις ε, μεταξύ τους ε, που τελικά η διαδικασία αυτή κινδυνεύει να γίνει απλώς μία, ένας ανθρωπιστικός διάβλος. Εν πάση ειλικρινία ε, μπορώ να σας πω ε, και πολύ φιλικά την άποψή μου. Ε, δηλαδή, εγώ δεν θέλω να κάνω γενικεύσεις. Υπάρχουν οπωσδήποτε κάποια ενδεχομένως στοιχεία ασαφή ακόμα και όχι αρκετά διαφανή και είμαστε φυσικά στη διάθεσή σας να τα συζητήσουμε. Αλλά παρόλα αυτά παραμένουν ε, οι ευθύνε ε, ε, και από πλευρά των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και πιστεύω ότι όσον αφορά την Μεσόγειο, το πρόβλημα δεν αφορά αυτούς που πάνε να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα νομικό, αφορά λοιπόν το τι γίνεται όταν έχουμε ανθρώπους που πρέπει να σώσουμε στις ακτέ τη Σικελίας ή στις ε, ακτές ε, γενικότερα ε, των νησιών της Ιταλίας. Το, το ζήτημα είναι νομικό και πρέπει να σας πω ότι ακόμα λύση δεν βλέπουμε και η απάντησή μας δεν είναι διαφρομένη. Εμείς εμείς σε όλες τις δημόσιες συζητήσεις καθημερινά λέμε ότι σταμάτησε ε, να έχει ε, έκτακτο χαρακτήρα ε, το θέμα της μετανάστευσης και έχει γίνει πλέον ένα φαινόμενο διαρθρωτικό και όχι συγκυριακό. εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω να σκέφτομαι ότι θα έχουμε μία Μεσόγειο με πλήθος βαρκών και πλοίων και δεν θα μπορούμε να δώσουμε μια λύση σε αυτό το διαφορετικό πλέον πρόβλημα. Ένα τρίτο ζήτημα, και θα ολοκληρώσω την παρέμβασή μου με αυτό, που συζητήθηκε πολύ και συζητήθηκε με κάποια σύμπτωση ε, απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων της ε, Ιταλίας και τον ε, κύριο Λόπος Αγγιλάρο, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας, είναι το θέμα το οποίο αφορά την ε, τροποποίηση της διαδικασίας ε, του Δουβλίνου. Εμείς συμφωνήσαμε και αυτή παραμένει ε, η Ιταλική θέση ότι υπάρχουν τρία κρίσιμα σημεία ε, τα οποία κατά την Ιταλική άποψη είναι δυσεπίλητα. Πρώτον, ε, η εισαγωγή μιας διαδικασίας η οποία δημιουργεί ακόμα περισσότερες περιπλοκές ε, παρά να λύνει ζητήματα. Δεύτερον, η ευθύνη της, ε, χώρας, ε, ε, της πρώτης χώρας άφηξης που γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη και τρίτον το θέμα της αλληλεγγύης. Η αλληλεγγύη είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, είτε είναι αλληλεγγύη είτε δεν είναι. Δεν είναι δυνατόν να επιχειρηματολογήσει κανείς για νομική αλληλεγγύη ή ανθρωπιστική αλληλεγγύη. Αυτά ήθελα να πω Πρόεδρε και σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ καλή η εισήγησή σας και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια, ε, έναν διάλογο με τους συναδέλφους. Αναφέρετε το ήδη τον κύριο Λόπετς Αγγιλάρ, την κυρία Τζουφρίντα. Ε, συνάδελφοι, ε, παρατηρήσεις, ερωτήσεις και κύριε Υπουργέ, στο τέλος, αν θέλετε, μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Χουάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ντομένικο Μαντσιόνε, μεγάλη μου χαρά σε ξαναβλέπω. Ήρθαμε εδώ. Θα, με, θα μιλήσω μετά ε, αγγλικά ε, αφού σε καλωσορίσω ε, και σε ευχαριστήσω για τη δέσμευσή σου και για την προσήλωσή σου σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο θέμα θέμα είναι εξαιρετικά επίπονο και σοβαρό ε, και αυτό το συμμερίζονται όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτήν την αποστολή. Ε, θα μιλήσω τώρα στα αγγλικά γιατί τα σημείο μου είναι ταγμένο στα αγγλικά. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη και κυρίως της αποστολής και κυρίως τις Ιταλικές αρχές ε, γιατί ήμασταν εκεί ε, Ήμασταν μια αντιπροσωπεία με μέλη ε, όλων των πολιτικών ομάδων ε, και αυτό για να δούμε μια κατάσταση που έπρεπε να την εξετάσουμε. Η εμπειρία μας ήταν ε, άκρος διαφωτιστική. Ήταν μια από τις πιο διαφωτιστικές μάλιστα στις οποίες έχω ε, συμμετάσχει ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το βασικό σημείο ήταν βέβαια η επαφή με τις αρμόδιες αρχές ε, για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης το μέτωπο, ας πούμε, γιατί είμαστε στα εξωτερικά σύνορα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Ιταλικά σύνορα είναι τα νησιά ε, και βέβαια τα hot spots. Θέλω να τονίσω την σημασία της ανταλλαγής ε, απόψεων που είχαμε, που ήταν εξαιρετικά μακροσκελής και εξονυχιστικές ε, μαζί με τους ε, εισαγγελείς, τους υπαλλήλους της στην Κατάνια. Ήταν εξαιρετική η επαφή και χαρήκαμε ε, ιδιαίτερως για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν όσον αφορά τις έρευνες που διεξάγουν οι Ιταλικές Αρχές και βεβαίως συμμερίζομαι την άποψη ότι η αλληλεγγύη χρειάζεται εδώ. Έχω επιμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της ε, συμμετοχής μου εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ότι η αλληλεγγύη δεν είναι πλέον ε, μια ε, ευχή απλά που διτυπώνουμε. Δεν έχει νόημα να βλέπουμε τόσα κράτη-μέλη εδώ απρόθυμα να δείξουν αλληλεγγύη στην Ιταλία ή στην Ελλάδα αλλά κυρίως στην Ιταλία γιατί ήταν προβλεπόμενη η κατάσταση που επικρατεί τώρα, ιδιαίτερα μετά από αυτή την υποτιθέμενη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τι σήμανε αυτό, ε, μια απλή παράκαμψη για το μεταναστευτικό κύμα, ε, για τους παράνομους διακινητές και τις μαφίες που περνάνε τον κόσμο από τη Μεσόγειο. Απλά αλλάξαν ρότα. Θέλω λοιπόν να μοιραστώ κάποιες παρατηρήσεις με τα μέλη της Επιτροπής. Ε, και καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω ε, ρητά την ευγνωμοσύνη μας προς την Ιταλική κυβέρνηση, προς τις υπηρεσίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στο Αγκούστο και στο Ποτσάλο για την επιτόπιση τη ε, προσφυγική κρίση στην Ιταλία. Και κατά δεύτερον, όλοι συμφωνούμε με την αξιολόγηση τη δύσκολη κατάσταση ε, σε ό,τι αφορά την ε, καταχώρηση τόσο πολλών μεταναστών και σε ό,τι αφορά στα σημεία εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε εντυπωσιασμένοι από τις θυσίες, από τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι Ιταλικές αρχές. Αλλά είναι προφανές ότι η νέα νομοθεσία για τους ασυνόδευτους ανηλίκους θα αποτελούσε ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι πραγματικά καταπήγον, δεδομένου του μεγάλου αριθμού ανηλίκων που καταφθάνουν. Πολλές τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν σημαντικές ε, περιορισμούς από πλευράς χρηματοδότησης. Όλες αυτές οι πολιτικές λιτότητας τι σημαίνουν στην πράξη. Ότι χώρες που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις αυτές, την πρώτη δηλαδή, βρίσκονται σε μια παράλογη κατάσταση που πρέπει να κάνουν τη δουλειά την οποία απαιτεί από αυτές ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως εξωτερικό σύνορο με πιο περιορισμένα μέσα και κονδύλια. Αυτό είναι παράδεκτο. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σε ό,τι αφορά και την ε, προσαρμογή της ε, νομοθεσίας και ο κανονισμός του Δουβλίνου προφανώς χρειάζεται να μεταρρυθμιστεί στα hot spots ε. ο εντοπισμός των προβλημάτων, το θέμα της ε, επανένωσης των οικογενειών, το δικαίωμα της οικογενειακής ζωής, η μεταφορά με αποτελεσματικό τρόπο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κράτηση ανηλίκων. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη κυδαιμονίας των παιδιών αυτών. Πρώτα λοιπόν τα παιδιά Και το θέμα της, ε, των αιτήσεων για άσυλο πρόκειται για κάτι παράλογο πραγματικά σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, απροθυμία των κρατών μελών να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν στο Συμβούλιο μέσα σε ψηφίσματα, σε συζητήσεις και μετά τα αρνούνται πάρα αυτά οι ίδιες οι κυβερνήσεις των κρατών μελών. Και τέλος, η ανάγκη μεγάλων αποστολών διάσωσης ε, και αναζήτησης ε, ατόμων. Η μεγάλη κλίμακα λοιπόν αυτή τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθούν ασφαλείς ε, και νόμιμοι οδοί εισόδου. Αυτό είναι ο τρόπος να δοθεί μία λύση σε όσους αναζητούν να μπουν στην Ευρώπη και τελικά καταλήγουν στα χέρια της μαφίας. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν ε, νόμιμοι εισόδου και το θέμα της επανεκατάστασης θα πρέπει να υπογραμμιστεί. Τα μέλη λοιπόν της αντιπροσωπείας καταλήγουν στο ότι η Ιταλία πλήττεται, πλήττεται βαριά από τη μάστιγα αυτή και αυτό θα έπρεπε να ξυπνήσει όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για όλη την ε, Ευρώπη, για κοινή αντιμετώπιση και αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, να ζητήσω από τους συναδέλφους που ήταν στην αντιπροσωπεία, ε, γιατί είναι μεγάλος ο κατάλογος των ομιλητών, αλλά να πάρει το λόγο η κυρία Σπινέλη, η οποία ήταν στην ε, αποστολική Κυριακή έγκαι Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα πρέπει να συμφωνήσω μαζί σας ότι με όλα αυτά που ακούσαμε από τους προηγούμενους ομιλητές ε, συμφωνώ. Συμφωνώ με τα πορίσματα, συμφωνώ με τα συμπεράσματα της συνεδρίασης μας στην Σικελία. να τονίσω ότι εγώ προσωπικά έχω εντυπωσιαστεί όλους ιδιαίτερους από την ε, δέσμευση που έχουν επιδείξει οι Ιταλικές αρχές και από την καλή διαχείριση της ε, μεταναστευτικής αυτής κατάστασης. Κατανοώ βέβαια ότι πήρε κάποιο χρόνο πρωτού βρεθούν στη θέση στην οποία βρίσκονται πλέον. Κάθε καινούργια άφηξη στην Ιταλία καταχωρίζεται πλέον και αυτό αποτελεί θεωρώ μεγάλο επιτεύγμα. Τώρα, να προσθέσω τρεις ερωτήσεις αν θέλετε στα σχόλια των προηγούμενων ομιλητών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τακτικά το σκέφτομαι μετά την επίσκεψή μας. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με το νομικό σκέλος, αν θέλετε το UNHCR, την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, κατηγόρησαν ότι είναι νομοθεσία θα περιορίσει τη διαδικασία για την χορήγηση του καθεστώτος ε, του πρόσφυγα και ότι θα περιορίσει τα δικαιώματα των ετούντων. Γιατί τα δικαστήρια ουσιαστικά χρησιμοποιούν μόνο μαγνητοσκοπημένα μηνύματα και δεν ακούν, δεν υπάρχει ακρόαση κανονική του ετούντα. Ως εκ τούτου θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι ακριβώς γίνεται τα δικαιώματα των ετούντων άσυλο, των ετούντων διεθνούς προστασίας, ε, διεθνής προστασίας εμ, παραβιάζονται γιατί καταλαβαίνω ότι χρειάζεται μια ταχύτητα στην ε, εκπαιρέωση των διαδικασιών. Από την άλλη όμως ε, υπάρχουν και τα πρότυπα και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεύτερη ερώτηση. η οποία σχετίζεται με τη συνεργασία των κυβερνητικών υπηρεσιών με τις ΜΚΙΟ. Σε πολλά επίπεδα είδαμε ότι είναι εξαιρετική η συνεργασία αυτή. Τοπικές και εθνικές αρχές, ιταλικές αρχές με, τα, με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Είναι τεράστιο το επίτευγμα αυτό και σας συγχαίρω. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως πώς γίνεται να βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου υπάρχει νομική αγωγή κατά μικείο η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για μία μικείο η οποία επίσης προσπαθεί να βοηθήσει την κατάσταση. Πώς είναι δυνατόν να μην μπορείτε να συνεργαστείτε για το θέμα αυτό. Προκειμένου να αποτελεί και υπόδειγμα, αν θέλετε, η Ιταλία. Παράδειγμα προς ε, μίμηση. Και αυτό σε ό,τι αφορά χώρες οι οποίες ε, αρνούνται να δεχτούν για παράδειγμα τους μετανάστες. Ερωτώ λοιπόν, γιατί δεν μπορείτε να συνεργαστείτε με καλύτερο τρόπο και πρέπει τελικά να καταφύγετε σε δικαστικές αγωγές. Τελευταίο ερώτημα. Αφενός ε, συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές σε ό,τι αφορά το σωστό επίπεδο άμα Και δεν είναι σωστό ότι κάποιες χώρες αρνούνται την μετεγκατάσταση. Θα έπρεπε κανείς να αναζητήσει κάποια λύση για το θέμα αυτό. Από την άλλη, μετά την επίσκεψη αυτή, πρέπει να πω ότι έχω την εντύπωση ότι η διαδικασία στην Ιταλία επιτόπου διαδικασία εννοώ για την μετεκατάσταση είναι τέτοια που τελικά είναι δύσκολη, βαριά και τελικά δεν γίνεται αυτή η μετεκατάσταση των προσφύγων. Πού βρίσκεται λοιπόν το πρόβλημα, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, στην πλευρά των άλλων χωρών, οι οποίοι υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υποδέχονται τα άτομα αυτά, ή μήπω το πρόβλημα προέρχεται από την ίδια τη διαδικασία και από τα εμπόδια που τίθενται σε τοπικό επίπεδο. Και εντάξει, για το δουλειά τα ακούσαμε ήδη. Ευχαριστώ, κύριε Σπινέλη. Eh, Ευχαριστώ κύριε Μαντσιόνε για την ε, παρουσίαση και κυρίως για τις τελευταίες ε, παρατηρήσεις όσον αφορά την ε, ευέλικτη αλληλεγγύη και το Δουβλίνο. Εγώ θέλω αν μου επιτρέπετε, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τη γραμματεία της Επιτροπής μας για την εξαιρετική, εξαιρετική έκθεση που συνέταξε όσον αφορά την αποστολή μας. Θα ήθελα δε να μιλήσω για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που εν μέρη ήδη αναφέρθηκαν από τη συνάδελφο το θέμα των ΜΚΟ, για τις οποίες έγινε πολλής λόγος και στην Ιταλία, όχι μόνο με τον ε, εισαγγελέα Τζούκαρο της ε, Κατάνια, αλλά και με τις ίδιες της ε, ΜΚΙΟ. Δεν θα ήθελα να θεωρηθούν οι δραστηριότητες των ΜΚΟ ως δραστηριότητες που μπορεί να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο ανθρωπιστικό διάβλο όπως είπατε κύριε Μαντσιόνε, γιατί κατά κάποιο τρόπο, κατά τη γνώμη μου, παρισφρεί επικινδύνωση η ιδέα ότι υπάρχει μια νέα αντίληψη νόμιμη στην Ιταλία και στην Ένωση που αποκαλείται έρευνα και διάσωση αλλά παράνομη. Γιατί η έρευνα και η διάσωση αφ' αυτού της είναι νόμιμη είναι νόμιμη εξορισμού, όπως και η ευέλικτη αλληλεγγύη. Αυτός ο όρος ευέλικτη αλληλεγγύη δεν στέκει, δεν πάνε αυτές οι δύο λέξεις μαζί. Έχουν γίνει λοιπόν, έχουν υπάρξει υπενιγμοί για τη ΜΚΟ, θα δούμε τα αποτελέσματα της ε, έρευνας, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία απτή απόδειξη. Όπως ε, δήλωσε και ο ίδιος ο υπεύθυνο της ε, οικονομικής αστυνομίας μας. Επίσης, ε, δεν θα ήθελα να γίνεται αναφορά στη μαφία όταν δεν έχουμε αποδείξεις, αν και οι εισαγγελείς μας έχουν τεράστια εμπειρία ε, για τα θέματα περί μαφίας. Κάτι ακόμα το οποίο είναι σημαντικό που αφορά την αποστολή είναι ο νέος Ιταλικός νόμος αντιπαράθεση στην παράνομη μετανάστευση και η συνάδελφος Μπάρμπαρα είπε πολύ σωστά πράγματα γιατί επικρατούν πολλές αμφιβολίες για αυτό το νομοθέτημα και για το κατά πόσο στέκει συνταγματικά τόσο γιατί αφορά τον αποκλεισμό άμεσης επαφής ανάμεσα στον κατηγορούμενο και στο δικαστή, δηλαδή η μαγνητοσκόπηση των επαφών, αλλά και ε, όσον αφορά την εφαρμογή της, των αποφάσεων, πράγμα το οποίο αμφισβητεί σύμφωνα με πολλούς ε, συνταγματολόγους αμφισβητεί την ισότητα των ε, πολιτών ενώπιον του νόμου. Τελευταία παρατήρηση για τις ΜΚΟ στην Ιταλία αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους. Πρόκειται για την νόμο Τζάμπα. Αυτός ο νόμος ήταν αντικείμενο επεξεργασίας κατόπιν τεράστια συνεργασίας ανάμεσα στις ΜΚΟ. Είναι μια, ένα εξαιρετικό νομοθέτημα. Τρίτη μου παρατήρηση είναι οι διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στην Ιταλία και τη Λιβύη. Συχνά έχουν επενεθεί αυτές οι συμφωνίες και εδώ σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ θέλω να σας μεταφέρω τα όσα άκουσα στην Ιταλία από τη ΣΜΚΙΟ και από την εκπρόσωπο της ε, είπα της του ΙΕ που υπογράμμισαν την φύση της Λιβύης ως παράγοντα όθησης. Δεν είναι πλέον μόνο χώρα διέλευσης, είναι μια χώρα από την οποία ο κόσμος προσπαθεί να ξεφύγει γιατί δεν υπάρχει κράτος και δεν σέβεται κανείς τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί. Έχουν ε, Μάλιστα, εκεί δημιουργηθεί τέτοιου είδους καταβλισμοί που αποκαλούνται στρατόπεδα συγκέντρωσης σας θυμίσω κύριε Μαντσιόνε ότι είναι παλιά ιστορία αυτή των συμφωνιών με τη Λιβύη γιατί το δικαστήριο του Στρασβουργού ήδη έχει καταδικάσει μια φορά την Ιταλία στην υπόθεση Λιέφη για την επαναπροώθηση προσφύγων από την Ιταλία προς την Λιβύη που ήταν επιστροφές μετά από τη συμφωνία ανάμεσα στον Περλουσκόνη και τον Καντάφη παλιά ιστορία λοιπόν η οποία χρονολογείται από την εποχή του Καντάφη και του Μπερλουσκόνη. Τέταρτη μου παρατήρηση, hot spot. Όντως, ε, ε, η αναγνώριση γίνεται και έχει φτάσει στο 100%. Υπάρχει και έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας που λέει ότι η αναγνώριση των προσφύγων θα πρέπει να γίνεται 100% αλλά ότι πολύ συχνά τα δακτυλικά αποτυπώματα καταφέρνουν να τα πάρουν ακόμα και συχνά με χρήση βίας. Ε, βέβαια η Ιταλία το αρνήθηκε αυτό αλλά η Διεθνή Σεμινιστή επιμένει. Τώρα όσον αφορά την μετεγκατάσταση για την οποία μπορούμε να πούμε ένα σωρό αρνητικά πράγματα αλλά που όμως κατά τη γνώμη μου, ε, γνώμη μου εάν δεν μεταρρυθμιστεί το Δουβλίνο η ίδια η μετακατάσταση αυτή η ιδέα είναι παραπλανητική. Και να σας δώσω μόνο ένα στοιχείο σε σχέση με την ε, Ιταλία. Το 2015 με 2016, ναι και κλείνω αμέσως Κλοντ. 2015 με 2016 στην Ιταλία μεταφέρθηκαν με βάση το Δουβλίνο, δηλαδή οι μετανάστες που φτάσαν στην Ιταλία πήγαν στην Ευρώπη και μετά επανεπιστράφηκαν προς την Ιταλία ήταν 5.000 τέτοιου είδους μεταφορές με βάση το Δουβλίνο και την ίδια χρονιά 3.936 μετεγκαταστάθηκαν. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι ξαναστέλνονται στην Ιταλία από αυτούς που μεταφέρονται από την Ιταλία. Εάν δεν υπάρξει μεταρρύθμιση του Δουβλίνου, η ίδια η επανεγκατάσταση κινδυνεύει να είναι παραπλανητική. Πρέπει να, να, να, εξυγχρονιστεί και πρέπει να δούμε τι προτείνει να κάνει, προτίθεται να κάνει η Ιταλική κυβέρνηση όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Σκοπεύει σοβαρά και πραγματικά να πιέσει για τη μεταρρύθμιση μέχρι ότου αυτή να ολοκληρωθεί στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ναι, πολύ καλή ερώτηση για το τι συμβαίνει με τις μετεγκαταστάσεις, επανεγκαταστάσεις και το Δουβλίνο. Ευχαριστώ συνάδελφοι, ξέρω ότι έχετε πολλά να πείτε όλοι, αλλά παρακαλώ δύο με τρία λεπτά ο καθένας για να προλάβουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις του Υπουργού. Επόμενη μιλήτρια η Σεσίλια Κέγγε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Κλόντ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό Μαντσιόνε για την συνθετική ε, εισήγηση που μας έκανε και για τη δική μας επίσκεψη. Και εγώ ήμουν ε, μέλος ε, της αποστολής αυτής και συμμερίζομαι τα όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα και κυρίως τα όσα είπε ο Χουάν Φερνάντο, γιατί ήταν μια αποστολή τόσο σημαντική που γιατί έτσι μπορέσαμε να δούμε επιτόπου αυτά που εμείς βλέπουμε μέσα στα βιβλία και τους νόμους, ε, τις ρυθμίσεις που συντάσσουμε. Το να πάμε επί τόπου, να δούμε με ποιο τρόπο λειτουργεί η ελληνική και να μπορέσουμε να Συνδυάσουμε όλες μας αυτές τις γνώσεις. Ήταν πολύ σημαντικό. Επισκεφθήκαμε τα hot spot, μιλήσαμε και για το θέμα των ΜΚΟ, αλλά και για τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Αλλά αυτό το κάναμε γύρω από ένα πολύ σημαντικό πυλώνα. Και εγώ από αυτό θέλω να ξεκινήσω, από την αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη που είδαμε με ποιο τρόπο μεταφράζεται σε, στην πράξη, επιτόπου. Βλέπουμε επίση ποια είναι η τεράστια προσπάθεια που καταβάλει η Ιταλία αυτή τη στιγμή. Το άρθρο 80 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει λόγο για αλληλεγγύη και για ίση κατανομή των ευθυνών, το λέει και από οικονομικής άποψης. Όταν όμως μεταβούμε επιτόπου, αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να τηρεί αυτό το άρθρο της ε, λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πόροι είναι πάντοτε λιγοστοί απέναντι σε ένα φαινόμενο που κάποιες στιγμές ε, παίρνει μορφή στιγμές-στιγμές ε, πολύ επίγουσες κατάστασης όπου ένα κράτος δεν μπορεί να φεθεί μόνο του. Όταν πρόκειται για τα hot spot και την ε, αναγνώριση, είδαμε όντως ότι έχει φτάσει το 100% αλλά δεν αρκεί η αναγνώριση και η ταυτοποίηση. Χρειάζεται η έρευνα και η διάσωση. Πρώτα απ' όλα να σώζονται οι ανθρώπινες ζωές. Εξετάσαμε και το θέμα των ε, ΜΚΟ. Το πρόβλημα δεν ισχύει μόνο στην Ιταλία. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν νέοι κανόνες, νέοι κανόνες πέρα από τους διεθνείς που μπορούν να εγγυηθούν τη λειτουργία των ΜΚΟ την ορθή λειτουργία των ΜΚΟ, αλλά και όλων όσων ασχολούνται με, αυτήν, ε, με αυτό το, το πρόβλημα της Μεσογείου και καλύπτουν στην ουσία το κενό της πολιτικής. Επίσης να εκφράσω την μεγάλη μου χαρά για το γεγονός ότι ως ε, Ευρωπαίο ε, πολίτη για φέτος τον ψαρά τον ψαρά από τη Ματζάρα Ντελβάλο. Αυτός ο άνθρωπος που έσωσε τόσες ζωές και είναι άνθρωποι μόνοι, μεμονωμένοι που καλύπτουν τα κενά και χρειάζονται περισσότερη προστασία και όχι να δέχονται επιθέσεις από πάνω. Επίσης για το Δουβλίνο θα πρέπει να ε, καθησυχάσω κύριε Υφυπουργέ ότι οι δικές μας εργασίες κατευθύνονται προς την ε, ε, αυτή την κατεύθυνση που αναφέρατε και εμείς στην Ιταλία ασχοληθήκαμε και με την, με την κατάσταση. Πήγαμε και επισκεφθήκαμε τα κέντρα υποδοχής αυτών των ανθρώπων και είδαμε πώς από εκεί ξεκινά η υπόθεση. Η κρίση της αλληλεγγύης, το γεγονό δηλαδή ότι πολλά κράτη-μέλη δεν θέλουν καν να υποδεχτούν κανέναν, επιλέγουν ποιου θα υποδεχτούν. Το συζητήσαμε, γυναίκες με παιδιά που εγκαταλείπονται εκεί. Τα κράτη-μέλη θέλουν ε, να διαλέγουν ό,τι τους βολεύει. Ακόμα και ενώπιον ανθρώπων που ανταποκρίνονται σε όλα τα κριτήριά μας. Αυτό εμείς πρέπει να το καταγγείλουμε και να το καταγγείλουμε έντονα. Γιατί αυτή η κρίση αλληλεγγύης δεν οδήγησε ακριβώς στην δυνατότητα ανταπόκρισης σε αυτή τη δράση αλληλεγγύης αυτής της πρότασης για κατάσταση. Αυτά όλα έχουν γονατίσει την Ιταλία και την Ελλάδα. Οι προσπάθειες λοιπόν που γίνονται επί τόπου μαζί με τις αρχές θα πρέπει να στηριχθεί αλλά και να ε, συμπληρωθεί γιατί πρόκειται για μια ε, γενική προσπάθεια ανάμεσα στους, ε, τους θεσμούς χρειάζονται πιο ισχυρές νομοθεσίες και εξωτερική πολιτική που θα ανταποκριθεί στα αιτήματα του Κοινοβουλίου, δηλαδή μια καθολική προσέγγιση, δηλαδή με σοδή, αλλά και δυνατότητα ανταπόκρισης στα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης. Να κλείσω λέγοντας ότι για μένα αυτή η αποστολή ήταν πολύ ουσιαστική. Έχουμε και για τους μη ασυνόδευτους ανήλικες, αλλά και για τις γυναίκες. Εμπόριο, εμπόρια των γυναικών. Να δούμε πώς οι γυναίκες μπορούν να ενσωματωθούν στο εσωτερικό της χώρας υποδοχής τους, κυρίως όσον αφορά την καταπολέμηση του εμπορίου ανθρώπων. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μαντζόνη που ήρθατε εδώ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ καλά οργανωμένη ε, από τη δική σας πλευρά αποστολή, αλλά να ευχαριστήσω και τη γραμματεία της Επιτροπής μας ε, ΛΥΜΠΕ, γιατί όλα κύλησαν πολύ ομαλά. Ε, κάναμε και κάποιες συναντήσεις με εισαγγελείς, με πολίτες, με τους δημάρχους των πόλεων κτλ. Και είχαμε την δυνατότητα να διαπιστώσουμε πολλά. Μας εξέπληξε η καλή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών. Πραγματικά είδαμε ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας, ιδίω δε ε, τα γραφεία της ε, ε, Frontex, όπου διαπιστώσαμε την πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των δυνάμεων των διαφόρων χωρών. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν πραγματικά πλούσιες οι εμπειρίες που αποκομίσαμε, κυρίως δε όταν πήγαμε στα hot spots. Okay, Καθώς επίσης και στο λιμάνι, το οποίο επισκεφθήκαμε. βλέπουμε ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη οι άνθρωποι αυτοί. Λέει ο κύριος Κρυπέκ. Βρίσκονται υπό διακριτική αστυνομική επιμέλεια κατά κάποιο τρόπο. Ε, και είδαμε ότι και οι διαταγές προστασίας εκδίδονται επιτόπου τόπου από εσά Μάθαμε, και αυτό μας εξέπληξε επίσης, ε, ότι μάθαμε λέω ότι ο αριθμός αφήξεων στο Ποτζάλο αφορούν ανθρώπους από τον Παγκλεντές και την Ιγυρία. Ε, ε, υπάρχει τεράστια διαφορά όμως σε σχέση με άλλες χώρες μέλη. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πόσο καλά γνωρίζουμε τι συμβαίνει στις χώρες αυτές γιατί ε, βλέπουμε ότι έρχονται και πολίτες ας πούμε από 30 διαφορετικές ε, χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Και διαπιστώσαμε λοιπόν ότι ε, υπάρχουν ένα στους πέντε είναι Πακιστανοί. Έχει αλλάξει λίγο και η ροή ε, των ανθρώπων που προέρχονται από την Ασία. Οι χώρες από τις οποίες προέρχονται έχουν αλλάξει. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί τροφή για σκέψη. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ε, να εστιάσουμε την προσοχή μας λοιπόν στα νέα αυτά στοιχεία. Το, στο Καστανόβο, η νέα, αυτό το κέντρο υποδοχής Ε, βλέπουμε, είδαμε μαθήματα γραφής και ανάγνωσης. Παρέχονται δε και άλλες υπηρεσίες. Και όλες οι υπηρεσίες είναι υψηλού επίπεδου. Μάθαμε όμως ότι ίσως κλείσει το κέντρο αυτό και αναφερθήκατε κι εσείς ε, ε, πλέον στην υπόθεση και στο φαινόμενο αυτό ως διαφορετικό και όχι συγκυριακό πλέον φαινόμενο. Ε, ε, υποψιάζεστε να έχει εμπλακεί η μαφία σε όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ακούσαμε εμείς ε, ότι, και ξέρουμε άλλωστε και τι λέει το ρητό, ότι τα φύλλα δεν κουνιούνται παρά μόνο εάν υπάρχει άνεμος, δηλαδή δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Ε, είδαμε Είδαμε ότι ακούσαμε μάλλον πάρα πολλά για λαθροδιακινητές, για μαφία. Ε, πρέπει να τα δούμε αυτά. Ε, πριν ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο η κατάσταση. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι εδώ παίζονται και πάρα πολλά χρήματα και από πλευρά της χώρας σας και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. υπάρχει, να μην το λησμονούμε αυτό, και ο εντός εγωγικών παράγων Λιβύη. Είδαμε και ανθρώπους, ε, εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων που μας έδωσαν μαγνητοσκοπημένο υλικό για τις φρικαλαιότητες ε, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στη, εκεί. Τέλος αναγνωρίζουμε ότι είναι τεράστιο το βάρος, το άχθος το οποίο καλείται να σηκώσει η χώρα σας. Και πραγματικά εξεπλάγιμε με θετικά όταν είδαμε πόσο καλά οργανωμένα είναι όλα αυτά τα πράγματα εκεί. Αλλά βλέπουμε ότι η οδός της Μεσογείου ε, μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Επόμενο ομιλητή, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερω, λέει ο κύριο Πολιέζε, τον ε, ε, υφυπουργό Μαντζιόνε και βεβαίω να ευχαριστήσω τον κύριο Λόπε Αγγελάρα αλλά και την Μπάρμπαρα ε, που, έχουν, που είχαν ηγηθεί τη αποστολή μα στην Ιταλία και του ευχαριστώ και για τα όσα μα είπαν σήμερα και την αναφορά που έκανα σήμερα ενώπιον μα. Πιστεύω ότι ήταν ιδιαίτερα ουσιώδη και σημαντική αποστολή και για τους ε, ε, Ιταλούς ε, που όμως δεν προέρχονται από την Σικελία αποτέλεσε και μια καλή ευκαιρία για να δούμε τα πράγματα στην πραγματικότητα, στην πραγματική ζωή γιατί είναι τόσο περίπλοκο το ζήτημα που είναι σημαντικό να βλέπουμε πώς ανταποκρινόμαστε σε αυτό. Να σας πω ότι από τη Ρακούσα και από τη Σιρακούσα από τις επαρχικές περιφερειακές σε αρχές ε, ε, μας ε, είπαν ότι, και αυτό το λέω και σε σχέση με την, με την συμφωνία με την Ιταλία, και μας είπαν ότι 5% των αποβεβαζομένων προέρχονται μόνο από την Σύρια. Από την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι καταλαβαίνετε ότι αυτό οδήγησε και στην αποτυχία του προγράμματος μετεγκατάσταση. Ε, και ε, επίσης γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι βάσει του κανονισμού η μετεγκατάσταση ε, γίνεται βάσει συγκεκριμένων αρχών. Ε, και επομένως αυτό το θέμα που είναι όνειδος ε, της μετεγκατάστασης, η κατάσταση δηλαδή αυτή η οποία δεν έχει προχωρήσει, καθορίζεται και από τις ιταλικές ροές οι οποίες είναι διαφορετικές και περιλαμβάνουν διαφορετικούς, διαφορετικούς μετανάστες από ότι η οδός των Βαλκανίων. Οπωσδήποτε θα πρέπει να τροποποιηθεί το Δουβλίνο 3 και ελπίζω ότι όλα τα κράτη-μέλη θα δείξουν ε, στάση ευθύνης και θα τροποποιήσουν ριζικά ε, το Δουβλίνο. Ε, Τώρα, η, ε, ε, το, το, διάταγμα ε, μηνύτη και σας μιλάω ως εκπρόσωπος της δεξιάς, νομίζω, νομίζω ότι πραγματικά ανταποκρίνεται, απαντάει σε μία εγγενή ανομαλία του Ιταλικού συστήματος που περιλαμβάνει ιδιαίτερα μακρές και χρονοβόρες διαδικασίες, διαδικασίες οι οποίες πρέπει να περάσουν από, από τους επάρχους, από τους περιφερειακούς, τα ε, κτλ. Και ε, γι' αυτό ε, οδηγούμε θα σε περιόδου ιδιαίτερα μεγάλες με ανθρώπου να μένουν μπλοκαρισμένοι στην Ιταλία για τρία και πάνω χρόνια. τώρα, οι νέε διαδικασίε βάσει και του σχετικού αυτού διατάγματο που ανέφερα προηγουμένω, όπου ε, στου τέσσερι μήνε ορίζεται η μέγιστη διάρκεια ε, τη αντιμετώπιση τη εξέταση τη έφεση, είναι κάτι θετικό. Τώρα, αυτό που θέλω να πω και τελειώνω είναι ότι ...4,6 δις ε, ευρώ είναι η πρόβλεψη για την επόμενη χρονιά... ...βάσει των στοιχείων που έχω στα χέρια μου ε, για την, ε, το κόστος που καλείται να σηκώσει το οικονομικό η Ιταλία... ...σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. λέει η κυρία Κινίτσι και εγώ θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω την αντιπροσωπεία ε, και ε, να σας ευχαριστήσω όλους αγαπητοί συνάδελφοι, όλους όσοι συμμετείχατε σε αυτήν την αποστολή. Νομίζω και το ακούσαμε και από τους συναδέλφους νομίζω ότι κατέστη σαφής ε, η τεράστια προσπάθεια που το σύνολο της Ιταλίας αλλά ιδιαίτερως η Σικελία ε, ε, καταβάλει μια προσπάθεια τεράστια και η οποία έχει καλυφθεί και από το ε, διάταγμα το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως αλλά ε, και από τις νομοθετικές αποφάσεις που είχε πάρει η Ιταλία όσον αφορά ε, τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Η Ιταλία ιδιαίτερος για το θέμα των νέων και των ασυνόδευτων ανηλίκων έκανε πάρα πολλά οι τοπικές αρχές, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι ίδιοι οι πολίτες ε, έδειξαν τον καλύτερο εαυτό τους, ε, έδειξαν στους ανήλικους και στους ασυνόδευτους ανήλικους ε, την απαραίτητη φιλοξενία και επιμέλεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους οι οποίοι πραγματικά μας μίλησαν για αυτή την πραγματικότητα την οποία εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, Καλά είπατε κύριε Υπουργέ ότι το θέμα της ε, μετανάστευσης ε, ε, αποτελεί πλέον ανθρωπιστική κρίση η οποία χρήζει δομημένης αλλά και δομικής αντιμετώπισης. Στις ακτές της Σικελίας πλέον βρισκόμαστε σε ευρωπαϊκά σύνορα και ως τέτοια θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι πρέπει, το είπαν και άλλοι και το λέω και εγώ, πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα του ασύλου. Είναι ε, αλήθεια ότι στην ουσία, όπως είπατε και εσείς, ε, αντί να βελτιώσει την κατάσταση, ε, χειροτερεύει η κατάσταση για τις χώρες της πρώτης υποδοχής. Και επομένως τα ίδια και τα ίδια και δεν αλλάζει τίποτα. Όσον αφορά την μεταρρύθμιση αυτή, πιστεύω ότι θα πρέπει κατά προτεραιότητα να ε, ληφθεί υπόψη η μεταρρύθμιση αυτή, γιατί πολύ καλά το είπε και ο συνάδελφος Αγγιλάρ. Ε, πρώτα απ' όλα μιλάμε για ε, παιδιά τα οποία είναι πρώτα παιδιά, έχουν πρώτα την ιδιότητα του παιδιού και μετά την ιδιότητα του μετανάστη επανειλημμένα από τους προλήσαντες συναδέλφους ε, αναφέρθηκε η λέξη αλληλεγγύη. Ναι, αλλά δεν χρειάζεται μόνο αλληλεγγύη, χρειάζεται και ευθύνη. Η υπευθυνότητα πρέπει να δείξουν όλες οι χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να αφήσουμε την Ιταλία μόνη της ή την Ελλάδα μόνη της. Όλες οι χώρες θα πρέπει να αναλάβουν ένα τμήμα της ευθύνης και ένα μέρος του βάρους και κατά την άποψή μου ε, και είναι σημαντικό και νομίζω ότι θα πρέπει να ε, κάνουμε περισσότερες προσπάθειες. Ε, θα πρέπει να να δημιουργήσουμε νομοθετικά εργαλεία συγκεκριμένα και πιο αποτελεσματικά όσον αφορά την αντιμετώπιση των μεταναστών. Λυπηρό θα ήταν εάν για να, δώσει, για να δώσουν όλη την συνεισφορά τους ε, όσον αφορά την ε, μετεγκατάσταση τη συνεισφορά τους λέω όλες ε, οι χώρες θα ήταν λυπηρό εάν ορισμένες χώρες αναλάμβαναν μόνο το φορτίο αυτό και όχι όλες μαζί να δείξουν ευθύνη και υπευθυνότητα. Η κυρία Αναγκόμες, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους που επένδυσαν τις Ιταλικές Αρχές και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που μετέβησαν στην ε, αποστολή. Την προηγούμενο Σάββατο ήμουν στο Σάντζου, στο σε ένα πλοίο που στα πλαίσια της αποστολής σε Σοφία δια, διαχειρίζεται τα υπόλοιπα πλοία της ε, αποστολής Σοφία στη Μάλτα μαζί με 11 μέλη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό που επιβεβαιώσαμε είναι ότι οι τελευταίες ε, ροές ε, ανθρώπων ήταν από τον Παγκλαντές, την Ιγυρία και το Μαρόκο. Αυτό μιλάει από μόνο του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει να αγνοεί στις εξελίξεις ε, την πολιτική και οικονομική πραγματικότητα στις χώρες αυτές, γιατί προφανώς αυτό επηρεάζει τι ροές των μεταναστών. Και φυσικά παληθεύσαμε ότι παρά τις κυβερνήσεις μας που βγαίνουν και λένε ότι είναι έτοιμες και προετοιμασμένες το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών εμείς το τραφοδοτούμε. Γιατί όσο του υπάρχουν νόμιμες οδοί, ελεγχόμενες οδοί άφηξης των ανθρώπων ως μετανάστες ως α, πρόσφυγες, εμείς τροφοδοτούμε την πίσνα. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Ό,τι και αν κάνουμε και έχει αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο, έχει προσαρμοστεί στις καταστάσεις και στα Βαλκάνια και στον τρόπο μεταφοράς Και φυσικά η Ιταλία, σύμφωνα με τις εκθέσεις, έχει ένα σύστημα νόμιμης άφηξης στο ανθρωπιστικό επίπεδο. Αυτό θα πρέπει να γίνει και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για να κλείσουμε πλέον την πίσνα των διακινητών. Αλλά δεν το κάνουμε αυτό γιατί, δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη όπως και είπε ο κύριος Μανσιώνα. Χωρίς αλληλεγγύη δεν γίνεται και ούτε το Δουβλίνο ούτε η μετεγκατάσταση δουλεύει. Δείτε για παράδειγμα την Πορτογαλία. Έχει λάβει τον τελευταίο χρόνο από την Ιταλία και την Ελλάδα χιλιάδες ε, πρόσφυγες. 40% των ανθρώπων αυτών που έχουν μετεγκατασταθεί έχουν φύγει μέσα σε ένα μήνα και λιγότερο, γιατί ήδη είχαν οργανωθεί να φύγουν να στους συγγενείς τους, εκεί που έχουν συγγενείς, στη Γερμανία κυρίως. Πολλοί πήραν τηλέφωνο να ευχαριστήσουν, αλλά τα είχαν όλα οργανωμένα από πριν και το παραδέχτηκαν. Όσο πιο πολύ χρόνο τους αφήνουμε στην Ιταλία και στην Ελλάδα, τόσο πιο πολύ χρόνο έχουν να οργανωθούν μέσω των ίδιων διακινητών. Και μετά τι γίνεται και με τους πραγματικούς πρόσφυγες από το Ιράκ, από τη Συρία. Αλλά αυτό δεν αποτελεί, αν θέλετε, το μεγαλύτερο τμήμα του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ιταλία. Έλαβα και αυτή την έκθεση χθες της ε, διεθνών προσφύγων που κάναν συνεντεύξεις με τον κόσμο στην Ιταλία και κατέληξαν ότι είναι φρικτή η κατάσταση στα hot spots και πρέπει να υπάρξει μια ειδική αποστολή και θα το προτείνω επίσημα για το τι συμβαίνει στα hot spots, τι συμβαίνει με τα παιδιά, τι συμβαίνει με τις γυναίκες θύματα σεξουαλικής βίας, βιασμού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Και δεν λαμβάνουν ούτε ιατρική, ούτε ψυχολογική βοήθεια στα hot spots. Ερώτηση προς εσάς κύριε Μαντσιώνα. Για την Λιβύα, εγώ είμαι κατά της εξωτερικής ανάθεσης των δικών μας ευθυνών και αρνούμε όπως αρνούμουν πάντα τη συμφωνία με την Τουρκία. Χθες από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήρθε μία προειδοποίηση για συλλογική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις μεταφορές από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Αλλά αυτό που με ανησυχεί επίσης πάρα πολύ είναι τα όσα συμβαίνουν με τη Λιβύη. Γιατί έχω επισκεφθεί τέτοια κέντρα κράτησης την εποχή του Καντάφη και του πολέμου και ξέρω ότι τα κέντρα αυτά κράτησης είναι ακόμα χειρότερα τώρα γιατί είναι σκλαβοπάζαρα, είναι στρατόπεδα βασανιστήριων. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιταλία τα ανέχεται αυτά με τη δικαιολογία ότι αναθέτουμε σε εξωτερικό παράγοντα τις ε, υποχρεώσεις μας, είμαστε υπέτη για την παραβίαση, τη φρικτή παραβίαση, κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα των μεταναστών στη Λιβύη μέχρι ότου υπάρξει κυβέρνηση στη Λιβύη και πολλά παραπάνω θα πρέπει να κάνουμε στη Λιβύη. Γιατί το θέμα δεν είναι η ασφάλεια στη θάλασσα. Είναι πραγματικά γελίο να γινόμαστε συνένοχοι με αυτά. Και να ρωτήσω, πόσοι, πόσοι τελικά επιστράφησαν από κράτη-μέλη όπως η Ιταλία, που είναι στην πρώτη γραμμή. Κώστα και Λόρεστον, συνάδελφοι, δύο-τρία λεπτά ο καθένας, για να έχουμε χρόνο να ακούσουμε και την απάντηση στα πολύ σημαντικά αυτά θέματα τα οποία θέσατε δώσω ερωτήσεις. Ο κύριος Κέστερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας και θα ήθελα να εκφράσω το σεβασμό που τρέφω προς την Ιταλική κυβέρνηση για τις ιδιαίτερες προσπάθειες που έχει καταβάλει για την ανθρωπιστική κρίση και την αντιμετώπιση της. Δύο ζητήματα θέλω να θέσω. Πρώτο, εξακολουθεί να είναι η κατάσταση η εξή. Πνίγεται ο κόσμο στο Μεσόγειο, πνίγονται οι μετανάστε. 1600 ω τώρα. Υπάρχει το πρόγραμμα τη Ιταλική κυβέρνηση Μάρεν το οποίο δεν συνεχίστηκε τόσο πολύ λόγω έλλειψης αλληλεγγύης ε, με τις Ιταλικές ε, υπηρεσίες και αρχές. Ε, ξέρω ότι προσπαθείτε να διασώσετε πάρα πολλά άτομα. Πόσοι περίπου μπορείτε να μας πείτε πόσους έχετε διασώσει με τις επιχειρήσεις αυτές και εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης συστηματικής, υποστήριξης πανευρωπαϊκά από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για υπηρεσίε για αποστολές διάσωσης, για να σταματήσει αυτή η ανθρώπινη τραγωδία που πνίγεται ο κοσμάκη στη Μεσόγειο. Να πάρει ένα τέρμα αυτή η κατάσταση. Όλε αυτέ οι ζωέ που χάνονται α, στη Μεσόγειο, γιατί τελικά έχουμε αρχίσει και συνηθίζουμε κιόλα. Να σα το πω και έτσι, το 2015 που πνιγόταν ο κόσμο σε Λαμπεδούζα, κάναμε και ενό λεπτού σιγή. Τώρα δεν θα είναι τόσο πολλοί κόσμο στη Μεσόγειο που δεν έχουμε καν χρόνο να τηρήσουμε ενό λεπτού σε γη. Βαθιά η καταστροφή και η τραγωδία. Και αν δεν κάνουμε κάτι, πολύ φοβάμαι ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσουμε να πείσουμε του πολίτε μα ότι α, σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεύτερο σκέλο τη ερωτήσή μου, το θέμα τη ευέλικτη αλληλεγγύη. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και μία άλλη, ένα άλλο σύστημα για να καλέσουμε τα κρατημέλη να δεχτούν μεταναστές. Ε, μήπως ένα σύστημα για κίνητρα θα μπορούσε να δουλέψει καλύτερα για τις περιφέρειες και για τις πόλεις για να μπορούν να υποδέχονται κόσμο. Ένα ενδεχόμενο ευρωπαϊκό ταμείο από το οποίο οι δήμοι και οι κοινότητες και οι περιφέρειες θα μπορούν να λαμβάνουν κονδύλια για να κάνουν επενδύσει σε κατοικίε, κοινωνικέ κατοικίε και το Αυτό θα βοηθούσε και τους πρόσφυγες, αλλά θα βοηθούσε και τον τόπιο πληθυσμό για να δημιουργηθούν θέσει εργασία κτλ. Μήπως να το και αυτό προκειμένου να υπάρχει καλύτερη κατανομή τελικά των προσφύγων. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τέλος, η Μάριον. Σας ευχαριστώ πολύ. Και συμφωνώ ιδιαίτερα με το θέμα που ακούσαμε για το ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο συντονισμένη βοήθεια από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε ό,τι αφορά όλους τους πόρους για να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα spots και καλύτερη αντιμετώπιση των παιδιών και των γυναίκων, αλλά όχι μόνο αυτών. Και τέλος, θα ήθελα να σας πω και το εξή. Όταν μας δίνετε αριθμητικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Ιταλία, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι από την Ελλάδα είναι πολύ πιο υψηλή, υψηλά τα ποσοστά της μετεγκατάστασης και από το Υπουργείο μας στην Εσθονία που πραγματικά εργά παρακολουθεί τα πράγματα και προσπαθεί να κάνει διάλογο με την Ελλάδα και την Ιταλία. Πρέπει να σας πούμε ότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Ελλάδα Έχουμε κόσμο που έρχεται από την Ελλάδα. Αλλά αυτό που ακούμε είναι ότι τα πράγματα στα hot spots ε, είναι πολύ πιο δύσκολα στην Ιταλία και είναι πολύ πιο δύσκολη η συνεργασία με, τα, με τις Ιταλικές αρχές και χρειάζεται πολύ πιο βαριά διαδικασία για τη με την μετεγκατάσταση και είπατε ότι αυτό κοστίζει η έλλειψη προετοιμασίας για τη μετεγκατάσταση. Το ερώτημα λοιπόν που έχω να θέσω είναι το εξή. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Η προθυμία των προσφύγων να προβούν σε την κατάσταση, οι πληροφορίε που του χορηγούνται, η συνεργασία με τα άλλα κρατεμέλη. Γιατί δεν είναι φυσιολογικό να παρουσιάζει η Ελλάδα τέτοιο βαθμό καλό συνεργασίας και όχι η Ιταλία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφοι για τις ουσιώδεις αυτές ερωτήσεις. Αν θα θέλετε παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να πάρετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλα τα ερωτήματα τα οποία άκουσα εδώ είναι σημαντικά. Ε, θα ομαδοποιήσω λίγο τις ε, απαντήσεις γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν συνάφεια λόγω περιεχομένου, λόγω θέματος κτλ. Όμως, εξ αρχής θα ήθελα να κάνω έτσι μία πρώτη προσωπική ε, σκέψη. Τέσσερα χρόνια εγώ έχω, είμαι στη θέση αυτή στο Υπουργείο Εσωτερικών και έχω σκεφτεί πολλά πράγματα, εξακολουθώ να έχω πολλές αμφιβολίες και ελάχιστες βεβαιότητες. Όμως έχω κάποιες βεβαιότητες. Πρώτον ότι η πολιτική που βλέπω ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η οποία θέλει να αντιμετωπίσει ένα θέμα το οποίο θα όφιλε να έχει όχι απλά ευρωπαϊκή αλλά ε, παγκόσμια διάσταση ε, ε, βλέπω ότι ε, αντιθέτως αφήνεται σε πολύ περιοριστικούς όρους και επομένως αποτελεί μια πολύ μεγάλη αποτυχία κατά την άποψή μου. Μια δεύτερη σκέψη ουσίας είναι η εξής, ότι όλοι στη συζήτηση αυτή επικεντρωθήκαμε στο θέμα της υποδοχής, ε, αλλά στην ουσία ε, η υποδοχή όπως και η διάσωση στη θάλασσα είναι ένα πρώτο βήμα μιας ε, πολύ μεγάλης πορείας την οποία οφείλουμε να κάνουμε όλοι μαζί. Γιατί τώρα να διασώσεις ανθρώπους και να μην ξέρεις μετά τι να τους κάνεις, πραγματικά είναι μια δραστηριότητα η οποία δημιουργεί απλά πρόβλημα στα εθνικά κράτη. Καθόλου απλό δεν είναι το θέμα και καθόλου δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μία χώρα μόνη της. Το 2015 έφτασαν, αποβεβάστηκαν διαθαλάσσεις 170.000 ε, άνθρωποι. Το 2016 181.000. Μέχρι σήμερα 61.000 ε, για το 2017, ε, που είναι κατά πολύ υψηλότερος αριθμός από την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς. Εμείς ε, λοιπόν ε, αντιμετωπίζουμε αυτά τα στοιχεία σαν να είναι απλά αριθμητικά στοιχεία, αλλά πίσω από τα αριθμητικά στοιχεία κρύβονται άνθρωποι ε, και που διαφέρουν και μεταξύ τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταξιδέψει με καλό τρόπο, ε, άλλοι οι οποίοι δεν ε, καταφέρνουν να φτάσουν στην ακτή και θάβονται, μένουν θαμμένοι σε αυτό το τεράστιο κημητήριο που είναι ε, η ε, Μεσόγειος. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι υφίστανται ε, ε, βιασμούς και κάθε άλλη μορφή σε βία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Δεν μπορούμε να του βάλουμε όλους σε ένα τσουβάλι λοιπόν. Απέναντι λοιπόν σε μια κατάσταση, σε ένα σενάριο σαν αυτό που σας περιγράφω, ε, ε, νομίζω ότι είναι περισσότερο σημαντικό να υπογραμμίσει κανείς την αλληλεγγύη και όχι ε, τον έλεγχο και να δείχνει κανείς με το δάχτυλο κάποιες χώρες λέγοντας ότι υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις. Κοιτάξτε, όταν ξεκινήσαμε τις διαδικασίες υποδοχής στην Ιταλία, ε, είχαμε τη δυνατότητα να υποδεχτούμε 25 με 29 χιλιάδες ανθρώπους ε, και τώρα έχει οκταπλασιαστεί και, και παραπάνω ε, η δυνατότητα αυτή. Έχουμε δυνατότητα υποδοχής 180.000 ανθρώπων. Στόχος μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε μικρούς και, μικρά κέντρα τα οποία θα έχουν μία ε, ε, τριχοειδή εξάπλωση ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε προβλήματα και θέλουμε να προχωρήσουμε μέσα από διαδικασίες συνένεσης με τις εδαφικές οντότητες και όχι μέσω της επιβολής. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις 180.000 ανθρώπους οι οποίοι αποβιβάζονται στην επικράτειά σου, χρειάζεται τρόπος και χρειάζεται και χρόνος για να τους αντιμετωπίσεις. Τώρα απαντήσεις. Ο, hot Ε, σας ε, εξήγησα πώς ε, ε, κατανοούμε εμείς τα hot spots και είναι γεγονός ότι είχαμε κάποιες καταγγελίες σχετικά με την χρήση βίας ή κάποιας μορφής βίας. Να σας πω, οι Ιταλικές αρχές έχουν αρνηθεί την ύπαρξη τέτοιων συμβάντων. Εγώ μαζί σας μπορώ να κάνω αξιολόγηση ε, του περιεχομένου, γιατί το να λέει κανείς απλά ε, έγινε, συνέβη αυτό ε, και το καταγγέλει στην, η Amnesty International στην έκθεσή της, λέω δεν παρόδο ότι ποτέ δεν ήρθε σε επαφή με τις Ιταλικές αρχές η οργάνωση αυτή. Να σας πω ότι είναι μικρή η αξιοπιστία πρώτον γιατί αναφέρεται σε ανώνυμες πηγές. Δεύτερον, γιατί αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος ε, ε, ανώνυμα ε, καταγγέλει κάποιες πράξεις οι οποίες δικαστικά δεν έχουν ποτέ καταγγελθεί. Τρίτον, νομίζω ότι είναι δυσλειτουργικό και σε σχέση με το στόχο. Εγώ πολύ συχνά έχω πάει στα hot spots και ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται ε, την ταυτοποίηση. Αυτό βεβαίως ε, είναι ένα από τα παράδοξα που προκύπτουν από το ε, Δουβλίνο. Δεν θέλουν να εγγραφούν, δεν θέλουν να καταχωριστούν γιατί θέλουν να προχωρήσουν το ταξίδι τους. Αυτό το Δουβλίνο που λέγαμε πριν ότι πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε. Κατανοώ βεβαίως ε, ότι μπορεί να είναι υποχρεωτικό ε, η υποχρεωτική λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων, γιατί εκεί μπορεί να υπάρξει πίεση. Αλλά εάν κανείς αν κανείς δεν δεχτεί ε, την λήψη των δακτυλικών του αποτυπωμάτων στην ουσία ε, ε, υποχρεώνει τις αρχές να τον στείλουν στα κέντρα τα οποία είναι κέντρα ανθρώπων προς απέλαση. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν συμβεί, ε, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί να συμβούν διάφορα στα hot spots, αλλά σε γενικές γραμμές πρέπει να σας πω ότι έχοντας πάει πολλές φορές σε hot spots, ε, είμαι ήσυχος και πιστεύω ότι είναι άδικο ε, να καταγγέλει κανείς τα hot spots για, για μεμονωμένα περιστατικά και να μην λαμβάνει υπόψη του τη συνολική εικόνα η οποία είναι θετική. Επόμενο θέμα. Ε, υπάρχουν ε, δεν ε, υπάρχουν ε, παράνομες ε, διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Δεν υπάρχει η έννοια της παράνομης διάσωσης. Κοιτάξτε, και εδώ δεν υπάρχει περιθώριο για διαφορετική νομική αντιμετώπιση. Αυτό όμως που μπορούμε να αναρωτηθούμε γιατί εδώ όντως υπάρχουν κάποιες φαίες ζώνες όπου μπορεί κανείς ε, να πει πολλά πράγματα. Ε, αυτό που μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό θέμα μπορεί να είναι η διαφάνεια. Ε, σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε παρούσες μη κυβερνητικές οργανώσεις στο, στην διεύλο της Σικελίας που δεν έπρεπε να είναι εκεί ή που εν πάση περιπτώσει δεν είχαν τα δικαιολογητικά που έπρεπε. Ε, και επομένως αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων έκαναν κάποιες διαδικασίες διάσωσης ε, αλλά θα έπρεπε τους ανθρώπους που έχουν διασώσει να τους, ε, φτά, να τους ε, παίρνουν στο λιμάνι, όπου στο λιμάνι θα, πρέπει, θα έπρεπε να έχουν κάποιες δομές. Και δεν είχαν τις δομές. Στην ουσία δηλαδή η διαδικασία συντονισμού πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει. Γιατί το να διασώσει κάποιον και μετά με δικό σου μέσο και μετά να πρέπει να χρησιμοποιήσει ε, ε, το πολεμικό ναυτικό ε, ή τι εγκαταστάσει που ήδη υπάρχουν έτσι ώστε να του υποδεχτεί, αυτό σημαίνει ότι σπάει η αλυσίδα της, του, του συντονισμού πέρα από αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, γιατί το πρόβλημα, όπως είπα και επανέλαβα, δεν είναι το θέμα της διάσωσης. Εμείς το, την κάνουμε την διάσωση και ποτέ δεν πρόκειται ε, να την εγκαταλείψουμε. Το πρόβλημα είναι ε, πολιτικών διαστάσεων να καταλάβουμε ότι οποιοδήποτε Ενεργεί στην Μεσόγειο θα πρέπει να βρίσκεται όσο γίνεται πιο κοντά στον ασφαλή λιμένα. Τώρα, αναφέρθηκε το ενδεχόμενο ε, εγκληματικών οργανώσεων. Ναι, φυσικά. Ε, τα μεγάλα κέντρα ε, είναι αυτά τα οποία ε, αφήνουν περιθώριο για την εγκληματικότητα και δεν νομίζω ότι αυτό συνέβη μόνο στην Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες. Και είναι αλήθεια ότι όταν μιλάμε πλέον για μεγάλους αριθμούς ε, μεταναστών, ε, οπωσδήποτε και λαμβάνοντας υπόψη την ε, οικονομία κλίμακος, είναι γεγονός ότι λόγω του όγκου των ατόμων μπορεί να υπάρχουν ενδεχόμενα κακής χρήσης ας πούμε ε, των ε, χρημάτων αλλά ε, και επειδή το αναφέρατε πρέπει να σας πω ότι η χώρα μου 4,2 δις αν όχι περισσότερα χρήματα τα οποία αφορούν και μονάχα την υποδοχή. Τώρα τι να σας πω, όταν μιλάμε ε, για τα 4,2 δις που βάζει η Ιταλία και τα 5 εκατομμύρια που βάζει ή τα 50 εκατομμύρια συγγνώμη, που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε ε, για σύγκριση αριθμητικών στοιχείων καταλαβαίνετε ότι τα χρήματα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν καλύψει ούτε ένα ελάχιστο τμήμα της ε, διάσωσης ε, και των επιχειρήσεων Μαρενόστρουμ. Επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε για κακή χρήση των ε, κοινοτικών χρημάτων. Εγώ αναφέρθηκα προηγουμένως στους ελέγχους και πόσο σημαντική είναι αυτή, όπως σημαντική είναι και η πρόληψη μέσω ε, μηχανισμών συγκεκριμένων τυποποιημένων συμβάσεων έτσι ώστε ε, να ε, ξεπεραστούν κάποιες δυσκολίες και έτσι ώστε να αποκλειστούν άνθρωποι με κακές προθέσεις, ας το πούμε έτσι. Νομίζω ότι αυτό που θέλουμε εμείς είναι μία ε, μεγάλη εδαφική διασκόρπιση, ας πούμε, κατανομή, ε, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει καλός έλεγχος. Ο καλός έλεγχος, ο βέλτιστος έλεγχος δεν γίνεται από τους χωροφύλακες, γίνεται από την πραγματική διάθεση ε, αλληλεγγύης και από την πραγματική βούληση ε, να ε, υλοποιηθούν μικρής κλίμακας και συγκεκριμένης εδαφικής ε, προσέγγισης προγράμματα ασυνόδευτη ανηλίκη Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για την Ιταλία και είναι μία από, τη, ένας από τα πιο σημαντικά νομοθετήματα που εγκρίθηκαν σχετικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορώ να πω ότι ένα πραγματικό ευρωπαϊκό σχέδιο με αναφορά στην κατανομή των ανηλίκων δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα. Και ωστόσο, εγώ μπορώ να σας πω ότι μόνο πέρσι ε, είχαμε 26.000 ε, παιδιά, ανήλικους ασυνόδευτους που αποβιβάστηκαν και μέχρι σήμερα έχουμε στις καταβλισμούς υποδοχής γύρω στα 16.000 παιδιά. Το κόστος είναι τεράστιο, είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το κόστος των ενηλίκων που φιλοξενούνται εκεί. Και εδώ προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, αλλά πραγματικά θα χαιρόμασταν αντί για το άγρυπνο μάτι του ελέγχου για να που εξετάζει αν εφαρμόζουμε όλες τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε με αυτή την νομοθεσία να έχουμε και ένα χέρι βοήθειας και συνεργασίας γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούμε ελαφριά τη καρδία να το αντιμετωπίσουμε. Νόμιμη οδή, διμερή συμφωνία με τη Λιβύη και υποκαλούμενη εξωτερήκευση, ανάθεση σε τρίτους. Από εμά εξαρτάται. Οι συμφωνίες με τη Λιβύη μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές. Ναι, εξαρτάται από εμά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα βεβαίω είστε ελεύθεροι εσείς να την επικρίνετε, ε, ακόμα και εντόνως. Αλλά η ιδέα ότι για τα επόμενα 20 χρόνια, και παραλαμβάνω αυτό που είπα πριν, εμείς θα συνεχίσουμε με ένα σωρό βαρκάκια να πηγαίνουμε ερχόμαστε στη Μεσόγειο, δεν έχει νόημα. Δεν δεν είναι διαρθωτικός τρόπος αντιμετώπισης αυτός. Εάν θέλουμε να κάνουμε μια απλή ανάθεση στους τρίτους, εγώ πρώτος και καλύτερος θα σας πω ότι πολύ πολύ με προβληματίζει και έχω τεράστιες αφιβολίες για το ότι και αυτό είναι μια κατάλληλη απάντηση στο πρόβλημα. Αν όμως αντίθετα θέλουμε να φτιάξουμε και να προσγειωθούμε και, κάποιο, και επίσης ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να αποβιβάζουν γιατί στη θάλασσα χάνονται πολλές ζωές, και μίλησα με τον γενικό σας εκπρόσωπο ε, πριν από δύο μέρες μόλις. Εάν μπορέσουμε να έχουμε κάποιες δομές τις οποίες θα διαχειρίζονται οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, και από τις οποίες ενδεχομένως θα είναι δυνατόν να αναγνωρίσουμε και να κάνουμε μία μετεγκατάσταση, δηλαδή να δημιουργήσουμε νόμιμες οδούς από εκεί, από τη Λιβύη. Αυτά δεν τα διαχειρίζονται οι λιβυκές αρχές. Ε, αν κάτι τέτοιο πετύχαινε θα είχε θετικό αντίκτυπο. Πέρα από την συμφωνία δηλαδή με την ε, Λιβύη. Από την άλλη πλευρά, η ιδέα της ανάληψης ευθυνών δεν μπορεί να ισχύσει μόνο για την Ευρώπη. Θα πρέπει αυτό, την ανάληψη ευθυνών, να την κάνουν και οι αφρικανικές χώρες από τις οποίες φεύγουν οι ροές ή, περνάνε οι ροές. Αυτό ήταν και αντικείμενο του συνεδρίου που συγκλήθηκε στη Ρώμη πριν από μία εβδομάδα και θα συνεχιστεί την Ισία μετά. Επαναλαμβάνω λοιπόν, εάν θέλουμε να εξωτερικεύσουμε, κατανοώ και συμμερίζομαι απόλυτα όλους τους προβληματισμούς. Από την άλλη πλευρά, καθώς πριν αναφερόμασταν σε ένα πείραμα που κάνει η Ιταλία, ακριβώς είναι ένα πείραμα ε, με τις θρησκευτικές κοινότητες ε, στο Σάντο Ετζίδιο υπάρχουν ε, Σύριοι οι οποίοι θα φτάσουν ε, στους χίλιους και που έφτασαν μέσω ασφαλού οδού. Ε, ήρθαν δηλαδή κατευθείαν σε εμά. Από ό,τι φαίνεται αυτό το πείραμα βρίσκει άλλα κράτη-μέλη ε, που θέλουν να συμβάλλουν και να συνεργαστούν. Πρώτη η Γαλλία εξέφρασε ενδιαφέρον, αλλά ακριβώς ε, για να τα συνδυάσουμε όλα αυτά θα σας πω ότι εγώ προβληματίζομαι απέναντι στη δυνατότητα δημιουργίας νομίμων οδών εάν δεν υπάρξει και συντονισμός για τις παράνομες οδούς που ήδη υπάρχουν, γιατί υπάρχουν κοινωνικά, πολιτικά ζητήματα, οικονομικά προβλήματα. Φοβούμε όμως ότι τα δύο πράγματα τελικά δεν θα πρέπει να ε, έρθουν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους, πράγμα το οποίο πολύ φοβούμε ότι θα γίνει. Τώρα, η μετεγκατάσταση ήδη από τη γέννησή της ήταν ε, προβληματική. Γιατί έχει δίκιο η συνάδελφος που το έλεγε πριν. Ακριβώς. Ε, έχουν ε, το θέμα της μετεγκατάστασης αφορά εκείνους που έχουν αναγνωριστεί ως δικαιούχοι ασύλου. Αυτό, δεν, αυτό είναι σύμπτωμα μεγάλης, μεγάλης δυσπιστίας, γιατί εμφανίζεται αυτό το 75% σε αυτό το πλάνο. Γιατί κανένας από εμά δεν εμπιστεύεται την αναγνώριση, τον εντοπισμό του διπλανού κράτους. Δηλαδή χρειάζεται ένα τόσο υψηλό όριο ώστε δεν θα μετεγκατασταθεί ένας άνθρωπος που μάλλον στη διπλανή χώρα ή στη δική μας χώρα δεν θα είχε πάρει μάλλον το άλσιλο. Οι ε, Σύριοι και οι ε, πολίτες της Ερυθρέας μόνο δικαιούνται αυτή τη στιγμή το άσυλο. Για τους υπόλοιπους υπάρχει μια ελάχιστη πιθανότητα με την κατάσταση και όπως είπα γενετής αυτή η ιδέα ήταν πολύ περιοριστική. Αλλά αυτό ισχύει και για τις άλλες ε, πανεγκαταστάσεις, αυτές που έγιναν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα συνεργάζεται περισσότερο από την Ιταλία για τον ε, βάσιμο λόγο ότι οι επαναγκαταστημένοι από την Ελλάδα θα έπρεπε να είναι 120.000, από εμά θα έπρεπε να είναι 40.000, οπότε είναι πολύ το φυσιολογικό ότι αυτοί που έρχονται από την Ελλάδα είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που έρχονται από την Ιταλία. Είναι και μόνο, και μόνο θέμα αριθμών. Το γεγονός όμως ότι είναι ότι δεν πρέπει μόνο η Ιταλία να δίνει τι πληροφορίες, γιατί ακριβώς η επανεγκατάσταση γίνεται μέσω του κανόνα, των κανονισμών του Δουβλίνου. Άμα τη χώρα που θέλει ε, να κάνει κατάσταση μας δίνει μια ολόκληρη σελίδα να συμπληρώσουμε, είμαι υποχρεωμένο να τη συμπληρώσω. Ε, θα πρέπει λοιπόν όντως να ασχοληθούμε και με το Δουβλίνο και για αυτά τα ζητήματα, γιατί Εάν θέλουμε να γραφειοκρατικοποιήσουμε και το σύστημα της μετεγκατάστασης, ε, θα λειτουργήσει ακόμα λιγότερο. Άφησα τελευταίο το νόμο Μινίτη. γιατί αυτό το νομοθέτημα προέκυψε από την εξή ιδέα, να επιταχύνουμε όσο γίνεται περισσότερο το χρόνο μέσα στον οποίο ολοκληρώνεται μία αίτηση ασύλου, γιατί τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια ε, είναι πολύ μακρύ χρονικό διάστημα. Και δεν, νομι... δεν σκέφτομαι μόνο τα δικαιώματα του ανθρώπου που θα αναγνωριστεί ή όχι, σκέφτομαι και τη λειτουργικότητα του συστήματος. Γιατί άμα έχω έναν άνθρωπο πέντε χρόνια πριν να το αποφασίσω αν θα του δώσω το άσυλο ή όχι, ε, τότε πρέπει να φτιάξω και ένα σύστημα το οποίο θα είναι πραγματικά ικανό να διευρύνεται επάπειρον. Γιατί διαφορετικά για πέντε χρόνια... Ε, μετά δεν θα μπορούμε πλέον να το διαχειριστούμε αυτό το σύστημα. Άρα λοιπόν ε, σκεφτήκαμε ότι η ε, καταχώρηση δεν είναι αρκετή. Πρέπει να υπάρξει και η διάλεξη από την Επιτροπή και από τη Δικαιοσύνη και στη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας από την Επιτροπή θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μία μαγνητοσκόπηση που μετά θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει η δικαιοσύνη αλλά η δικαιοσύνη έχει το δικαίωμα να καλέσει και τον ενδιαφερόμενο, αν δεν τη αρκεί αυτή η μαγνητοσκόπηση. Οπότε πραγματικά ειλικρινά ο στόχος ήταν να συνδυάσουμε, μάλλον να επιτύχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα στην ε, ε, διεκπαιρέωση αυτής της διαδικασία χωρίς να επιβαρύνουμε ή να βλάψουμε τα δικαιώματα του ετούντος άσυλο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαντσιώνε. Σας ευχαριστώ συναδέλφοι αν θέλετε ε, να ευχαριστήσω τον Υπουργό, να ευχαριστήσω και τα μέλη που συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία αυτή, γιατί και για αυτή την αντιπροσωπεία και για την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα πραγματικά πιστεύω ότι οι βουλευτέ ενεπλάκησαν σε πολύ προσωπικό επίπεδο και όπω ε, βλέπετε ε, έχουν ασχοληθεί επισταμμένω με το φάκελο αυτό, για το Δουβλίνο, για την επενεγκατάσταση. Κάποιοι συνάδελφοι δεν μπορούσαν να είναι εδώ, αλλά έχουμε πραγματικά μεγάλη εμπειρία μεταξύ των βουλευτών. Να κατανοήσετε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη δέσμευση από δική μα πλευρά και χαιρόμαστε που μπορέσατε κι εσεί να έλθετε μετά την αντιπροσωπεία. Προφανώ πολλά πρέπει να κάνουμε. Ακόμα και σήμερα το απόγευμα, μάλιστα, συνεργόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα παιδιών και μετανάστευση. Είναι πραγματικά μεγάλη η δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να το έχετε υπόψη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας αφιερώσατε για την συζήτηση αυτή για πολύ ευαίσθητα ζητήματα και δυστυχώ είναι τόσο α, πυκνή ημερήσια διάταξη που δεν μπορούμε να σας αφιερώσουμε πιο πολύ χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και εσάς και τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ. So colleagues, Συνάδελφοι, να περάσουμε τώρα πάρα αυτά στην κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και με την Επιτροπή ΦΑΜ. Να ζητήσω από την Πρόεδρο της Επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών να έλθει εδώ στο Προεδρείο. Είναι μια σύντομη συνεδρίαση μισής ώρας. Να κάνω τα εισαγωγικά σχόλια σου καταφθάνει η Πρόεδρος.